στο τελευταίο. Buongiorno a tutti. Iniziamo i lavori di questa Λοιπόν, ξεκινάμε τις ε, εργασίες μας. Ε, υπάρχουν τα θέματα στην ημερήσια διάταξη, το αποτέλεσμα των εργασιών της συνεδρίασης των συντονιστών. Εχθές ε, οι συντονιστές αποφάσισαν για το θέμα που έχει σχέση με την διαδικασία, επαλήθευση της διαδικασίας την οποία είχαμε γκρίνει για να επιλέγουμε κάπως τις αναφορές έτσι ώστε η εργασία μας να είναι περισσότερο αποτελεσματική και αποφάσισαν να τηρήσουν την ε, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία αντέδρασε, διαφώνησε στη διαδικασία που είχαμε προτείνει εμείς και η οποία νομική υπηρεσία λοιπόν πρότεινε μια εναλλακτική διαδικασία και με αυτή τη διαδικασία θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Αυτή λοιπόν η εναλλακτική διαδικασία αφορά στο να αξιολογούνται, να υποβάλλεται αξιολόγηση του κατά πόσον είναι αποδεκτές ε, οι αναφορές ε, και αυτό θα, η απόφαση για αυτή την αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ε, οι ε, αναφέροντες θα ε, δέχονται λοιπόν αυτή την αξιολόγηση από τα μέλη και της δικής μας επιτροπής. Θα υπάρχει σε εσά, θα δείτε ένας κατάλογος όλων των αναφορών για τις οποίες αναφορές θα πρέπει να αποφαινόμαστε το μη παραδεκτό η επίτροποι βέβαια και οι διάφοροι άλλοι αρμόδιες επιτροπής ε, θα μπορούν επίσης να αποφαίνονται. Αυτή είναι η άποψη που επικράτησε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Εμείς θα καταθέσουμε αυτή την άποψη στη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διαπιστώσουμε κατά πόσον αυτή η απόφαση είναι συμβατή με τους ε, κανόνες ε, της συνθήκης και με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Άουκεν, θέλετε παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Μάλιστα. Νομίζω αυτό που είπατε είναι αποδεκτό, αλλά πρέπει να πούμε επίσης ότι δεν έχουμε καμία άλλη δυνατότητα. Να πούμε ότι ε, δεν είναι πολιτική απόφαση, ε, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ε, τηρήσουμε τη νομοθεσία και εάν ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η Νομική Υπηρεσία αποφαίνονται αυτό που αποφάνθηκαν, νομίζω ότι αυτό είναι αποδεκτό και πρέπει να αναζητήσετε έναν τρόπο για μια ταχεία διαδικασία. Βεβαίως ε, πρέπει να είμαστε αρμόδιοι, αλλά μια ταχεία διαδικασία για όλες τις ε, περιπτώσεις τις οποίες συζητήσαμε χτες. Οι διαδικασίες να μην είναι χρονοβόρες, αλλά να είμαστε ε, σίγουροι τουλάχιστον ότι λειτουργούμε νομότυπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Άουκεν. Το δεύτερο θέμα που ελήφθη υπόψη που συζητήθηκε ήταν η αναφορά σχετικά με την καταστροφή που έλαβε χώρα στο Σμόλενσκ. Επ' αυτού του σημείου η, Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή μας μάλλον ζήτησε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και η νομική υπηρεσία σε συμφωνία με το προηγούμενο θέμα μας ε, είπε ότι θα πρέπει να γίνει μια δήλωση παραδεκτού εκ μέρους της Επιτροπής. Ε, βέβαια ε, μόνο ε, πολιτικό όργανο μπορεί να αποφανθεί τελικά. Κατόπιν τούτου οι συντονιστές ε, αξιολόγησαν αυτήν την αναφορά και αποφάσισαν ότι αυτή είναι παραδεκτή και ε, μετέθεσαν για την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών για το πότε θα ενταχθεί αυτή η αναφορά στην ημερήσια διάταξη. Εξάλλου κατεπίγουσες ε, κρίθηκαν δύο αναφορές, ε, κυρίως ε, η αναφορά που έχει ως αντικείμενο τη Συμφωνία Άκτα και επίσης και η αναφορά που αφορά στο να ξεκινήσει μια διαδικασία σχετικά με μια νέα χωματερή που πρόκειται να κατασκευαστεί στο Λάτσιο στην Ιταλία οι συντονιστές ε, συζήτησαν ε, το αποτέλεσμα της ε, συνεδρίασης της πρώτης ομάδας εργασίας που αφορά στο νόμο περί των παράκτιων περιοχών στην Ισπανία και συζήτησαν επίσης το κατά πόσον θα πρέπει να σταλεί μια επιστολή στον Ισπανό αρμόδιο Υπουργό. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η απόφαση των Ισπανικών αρχών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω, όπως έγινε και χθε με τους ε, συντονιστές, ότι είχαμε μία συνάντηση κατά τη διάρκεια του Στρασβούργου με τον ε, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς. Και εγώ ε, συζήτησα με τον κύριο Σούλτς το θέμα, το πλέον, τα πλέον ευαίσθητα θέματα, τα θέματα με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή μας και τα θέματα τα οποία παρουσίασε και εκείνο όταν ανέλαβε το αξίωμα του Προέδρου. Το πρώτο θέμα έχει σχέση με την ε, μία και μόνη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό, αν θυμάστε, το έθιξε ο κ. Ε, κατά την τελετή ανάληψη των καθηκόντων του. Ε, έχουμε μία αναφορά σχετική που κατατέθηκε από πάνω από ένα εκατομμύριο αναφέροντες, πολίτες και υπάρχει και το θέμα της λαϊκής πρωτοβουλίας. Επ' αυτού λοιπόν παρουσίασα στον ε, κύριο Σούλτς ε, το θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για τον ενδεχόμενο ε, τροποποίησης των κανονισμών. Όλο αυτό το θέμα αφορά βέβαια το ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή μας. Ο πρόεδρος ε, κύριος ε, Σούλτς ε, στη δική του την ομιλία κατά την ε, τελετή ανάληψη ε, των ε, καθηκόντων του δεσμεύτηκε να μας στηρίξει στη συζητήση για αυτά τα δύο τόσο σημαντικά θέματα. Και όσον αφορά το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης εχθές αναφέρομαι στην οργάνωση των επισκέψεών μας σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εχθές λοιπόν διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά δεν αποφασίσαμε ακόμα για τις επισκέψεις που θα κάνουμε. Και οι χώρες οι οποίες, θα, οι επισκεφτήκαμε το 2011, αυτό που είχαμε αποφασίσει το 2011, βεβαίως και ε, επιβεβαιώθηκε και θα πρέπει απλά να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί. Επισκεφθήκαμε την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πολωνία και πρέπει να δούμε κατά πόσον ε, σε αυτές τις επισκέψεις ε, μπορούμε να προσθέσουμε και ε, μια άλλη χώρα που να έχει άμεση σχέση με ευαίσθητες αναφορές. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό το θέμα θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε διεξοδικά στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών, τότε να λάβουμε την τελική απόφαση και οι συντονιστές ε, ανέλαβαν τη δέσμευση να κάνουν μια συγκεκριμένη πρόταση στο Προεδρείο και κατόπιν το Προεδρείο και αυτό θα παρουσιάσει τη δική του άποψη στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Δεν έχω άλλα θέματα για να σας ε, αναφέρω ε, θέματα που να ετέθησαν στη διάρκεια της συνεδρίας των συντονιστών και δίνω το λόγο στον κύριο Γιάρ. Ευχαριστώ. <clears throat> Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για το θέμα της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών που εξακολουθείτε να επιμένετε για να αναγνωριστεί η αρμοδιότητα της ε, ε, Επιτροπής μας και φαίνεται να έχετε κάποιες πρώτες επιτυχίες με τις συνεργασίες με τον νέο Πρόεδρο. Και εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας. Συμφωνώ απολύτως. Αν μου επιτρέπετε να αναφέρω σχετικά στην παρούσα επιτροπή. Εγώ είμαι εισηγητή εδώ, αλλά είμαι και σκιώδη εισηγητή στην ΑΦΚΟ για θέματα συνταγματικά. Εκεί έχει κατατεθεί αίτηση έτσι ώστε να ρυθμιστεί το θέμα της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών ώστε η Επιτροπή Αναφορών να μην συμμετέχει. και επομένως να κρίνει η Προεδρία της ε, ε της ε, Ομάδας των Πρόεδρων των Επιτροπών ποια Επιτροπή θα λαμβάνει την αρμοδιότητα. Μετά από πολλές συζητήσεις προβλέπεται τώρα σε μία τροπολογία μετά από αίτηση της Επιτροπής Αναφορών η διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών να αποφασίζει εάν θα συμπεριλαμβάνονται και μονομένα μέλη της Επιτροπής Αναφορών. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες της παρούσας Επιτροπής και ούτε ανταποκρίνεται και στα όσα ομοφόνος έχουμε μέχρι τώρα συζητήσει στις διάφορες επιτροπές. Γι' αυτό εγώ έθεσα υπόψη της Συνταγματικής Επιτροπής και τα θέματα αυτά και διαπραγματεύομαι με τους συναδέλφους μου εκεί μια συμβιβαστική λύση. Για την ώρα πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό και εσείς, δηλαδή οι, και οι συνάδελφοί σας στις δικές σας πολιτικές ομάδες να συνεχίσουν να τηρούνται ενήμεροι. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί αυτό το νέο μέσον ή εργαλείο, αν θέλετε, του της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών και να μείνει εντελώς εκτός η Επιτροπή Αναφορών. Νομίζω λοιπόν πρέπει να γίνει παρέμβαση παρά το Προέδρο από κάθε δυνατή γωνία και πτυχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα ουσίας και αν κατάλαβα καλά μου υπενθυμίζετε ότι και την Παρασκευή εκπνέει διορία για την κατάθεση τροπολογιών. Ε, κατόπιν τούτου και εμείς ε, πρέπει να ε, καταθέσουμε τη δική μας την τροπολογία η οποία απλά επιβεβαιώνει την απόφαση που έχει ήδη ληφθεί κατά το παρελθόν. Η συνάδελφος κυρία Αούκεν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια για τις διερευνητικές επισκέψεις. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά δεν είναι θέμα διεξαγωγής επίσημων ε, συναντήσεων στις πρωτεύουσε. Ουσιαστικά εμείς τις αναφορές εξετάζουμε και παρακολουθούμε. Μπορεί να μην σας κατάλαβα καλά. Ελπίζω ότι δεν άλλαξε η διαδικασία που ακολουθούμε, δηλαδή ότι εμείς επισκεπτόμαστε περιοχές, ε, όχι δεν κάνουμε επίσημε επισκέψεις, δεν είναι αυτή η δουλειά μας, ε, ε, ξέρετε και πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνο μας. Δεν κάνουμε επίσημε επισκέψεις, επισκεπτόμαστε τις περιοχές για τις οποίες υπάρχει αναφορά. Να σας εξηγήσω λοιπόν. Οι τέσσερις ε, χώρες ε, τις οποίες ανέφερα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Πολωνία, οι χώρες αυτές επελέγησαν πέρυσι το 2011 ως ε, προορισμοί δική μας για θεσμικές επισκέψεις. Δηλαδή για να γνωρίσουμε επιτόπου την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες αυτές. Δεν είχαμε ούτε το χρόνο ούτε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτές τις επισκέψεις. Απλά λοιπόν εχθές επιβεβαιώσαμε ότι θέλουμε να πάμε σε αυτές τις χώρες και οι συντονιστές μετά από πρόταση ορισμένων ομάδων είπαν, πρότειναν όταν θα επισκεφτούμε τις χώρες αυτές να συνδυάσουμε την επίσκεψή μας και με την εξέταση κάποιων αναφορών που θα προέρχονται από τις χώρες αυτές. Κυρία Ουκεν, δεν νομίζω ότι ποτέ λάβαμε τέτοια απόφαση, δηλαδή ότι θα περνάμε το χρόνο μας στις πρωτεύουσε. Μα δεν έχουμε χρόνο. Δεν θα μπορέσουμε να επισκεπτούμε επιτόπου τις περιοχές που θέλουμε να δούμε. Για κοιτάξτε καλά την ημερήσια διάταξη της συνδρασίας των συντονιστών. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να πηγαίνουμε εκεί που υπάρχει αναφορά. Να δούμε αναφέροντες. Όταν ήμουν ε, στη Δανική Βουλή περνούσα ώρες και ώρες με επισκέψεις ε, ευγενία, αν θέλετε, επίσημες επισκέψεις. Όχι, δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να δουλεύουμε μαζί με τους αναφέροντες. Κοιτάξτε, πέρυσι λάβαμε μία απόφαση και χτες την επιβεβαιώσαμε. Και ως πρόεδρος σας είπα τι είπαμε χτες. Εσείς λέτε αυτό που είπατε, αλλά δεν μπορούμε κάθε φορά να αμφισβητούμε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Πέρυσι λοιπόν αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε επισκέψεις οι οποίες θα είναι πρόσθετες από αυτές που κάνουμε για να ασχοληθούμε με αναφορές. Ε, Βεβαίω, αν συμφωνεί οι αν θέλετε να αλλάξουμε την απόφασή μας. Γι' αυτό σας είπα τι είπαμε, τι αποφασίσαμε χθε το βράδυ. Μετά από πρόταση ορισμένων συντονιστών, αποφασίσαμε λοιπόν να ε, συνδυάζουμε τις επισκέψεις μας όταν επισκεπτόμαστε μια χώρα μαζί με, με την εξέταση των αναφορών. Ο συνάδελφος κύριος ε, Γιάρ έχει το λόγο. Κοιτάξτε, σωστά τα παρουσιάσατε κυρία Πρόεδρε και σας παρακαλώ πολύ κάποια ψυχραιμία, λίγη ψυχραιμία. Γιατί ε, πρέπει να πούμε το εξής, έχουμε πολλές ε, ε, και καλές ιδέες, αλλά για λόγους έλλειψης χρόνου και σύνθεση ομάδας δεν κατορθώνουμε να επιτύχουμε το στόχο της αποστολής. Ψυχραιμία λοιπόν. Ποτέ ε, δεν ακυρώθηκε μια επίσκεψη που ήταν σημαντική για μας. Κάθε άλλο, μερικές φορές αναβάλαμε, αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε επισκέψεις, είτε γιατί δεν είχαμε αρκετούς ε, ε, είτε δεν πετύχαμε σωστά θέματα στη μέση διάταξη. Ψυχραιμία λοιπόν, ε, το θέμα είναι να έχουμε βεβαιω μια καλή μερίσια διάταξη, αλλά είναι επίση σημαντικό να έρχονται και αρκετοί βουλευτέ ε, και να βρίσκουμε και κάποιο χρονικό διάστημα ή κάποια χρονική στιγμή που μα βολεύει. Δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση προσφέρεται για να ξεκινήσει τώρα πόλεμο, που δεν νομίζω ότι ενδείκνυται έτσι κι άλλιω Πρόεδρος. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλος το λόγο. Πάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η συνάλφος κυρία Μέρκης, θέλετε να μιλήσετε για το προηγούμενο θέμα. Παρακαλώ. Ναι. Δεν ξέρω αν σας κατάλαβα καλά. Αν έχω παρακολουθήσει τη συζήτηση τουλάχιστον. Βέβαια δεν ε, ήμουν παρούσα στην συνεδρίαση των συντονιστών, άρα δεν είχαμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε, αλλά τι ακριβώς μας προτείνεται τελικά να μην διενεργούμε ερευνητικέ επισκέψει γιατί δεν έχουμε χρόνο. Καλά κατάλαβα. Eh, Κοιτάξτε, δεν πρότεινα κάτι τέτοιο. Εγώ απλά σα μετέφερα αυτά που πρότειναν οι συντονιστέ. Δεν έτεχε θέμα να αντικαταστήσουμε τις αποστολές με επισκέψεις. Απλά προτάθηκε να παραμείνουμε πιστοί σε αυτό που αποφάσισαν πέρυσι οι συντονιστές. Και εγώ απλά σας το μετέφερα. Είπαμε να κάνουμε και επισκέψεις σε διάφορες χώρες. Και οι χώρες αυτές είναι οι τέσσερις που σας ανέφερα. Σύμφωνα λοιπόν με την πλειοψηφούσα άποψη των συντονιστών επιβεβαιώνονται αυτές οι τέσσερις χώρες. Δηλαδή, επιβεβαιώθηκε η απόφαση των συντονιστών της περσίνης χρονιάς. Το Προεδρείο απλά ε, μεταφέρει και επιβεβαιώνει την ε, απόφαση των συντονιστών. Τώρα, αν οι συντονιστέ ε, θέλουν να αλλάξουν μία απόφαση, η συνεδρίασή μας είναι κυρίαρχη και μπορεί να τεθεί εδώ το θέμα. Ο κύριος Μποστινάρου. Κυρία Πρόεδρε, είναι προφανές ότι οι επισκέψεις και οι διερευνητικές επισκέψεις διαφέρουν από τις άλλες επισκέψεις και θεσμικά και έχουν άλλη έννοια. Αλλά θεωρώ ότι όταν πηγαίνουμε σε μια χώρα είναι απαράδεκτο να μην ε, συναντώμεθα με τους ε, αναφέροντες και να μην βλέπουμε το γενικότερο πλαίσιο. Γιατί πηγαίνουμε σε αυτά τα κρατη τελικά. Είναι άχρηστο, εντελώ άχρηστο να μεταβούμε, παραδείγματο χάρη στην Πολωνία, όπου γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο λόγο τη επίσκεψή μα εκεί είναι αυτό το, αυτή η ανοιχτή πέθρια εκμετάλλευση ανθρακοριχείο ή να πάμε στην ε, Ισπανία ή οπουδήποτε άλλο ή στην Ιταλία. Γιατί πηγαίνουμε στην Ιταλία. Υποτίθεται ότι αυτό γινόταν σε συνέχεια της επίσκεψης στην Καμπανία. Άρα, για θυμοτυπικούς λόγους πηγαίνουμε από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Όχι, είναι άχρηστο κάτι τέτοιο. Καλύτερα να εξοικονομήσουμε τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μην κάνουμε τέτοια ταξίδια. Πρέπει να συγκεράσουμε και τις δύο πτυχές, δηλαδή στις επισκέψεις μας, ναι με να συναντώμεθα και με κάποιους ε, αξιωματούχους, αλλά και με τους αναφέροντες για να δείξουμε το δέοντα σεβασμό, την εκτίμηση προς τους πολίτες των κρατών μελών. Αλλιώς είμαι αντίθετος να γίνονται θυμοτυπικές επισκέψεις, να στείνεται και το κόκκινο χαλί για τους ε, βουλευτές. Όχι δεν έχει από πολιτικής πλευράς κανένα νόημα. Εγώ είμαι υπέρ να συνδυάσουμε τα δύο στοιχεία. Δηλαδή, ας έχουμε πιο σύντομο ε, πακέτο, αν θέλετε, επισκέψεων, αλλά να είμαστε αποτελεσματικοί και ως προς τη διερευνητική μας αποστολή. Όχι απλά να αποτείουμε φοροτιμή σε υπαλλήλου ή σε μέλη των κυβερνήσεών μας. Πολύ ωραία, συμφωνώ απόλυτα. Ε, με αυτό που είπατε και με αυτό που αποφάσισαν εχθές οι συντονιστές. Ας κλείσουμε αυτό το θέμα και ας περάσουμε στο επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης ε, που είναι η ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Ο συγητής είναι ο κύριος Σαλαβράκος. Κύριε Σαλαβράκο, θέλετε να λάβετε το λόγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. παρακαλώ. Θέλω να πω πολλά, το, το είχα αναπτύξει. Ε, έχω δεχθεί όλες τις τροπολογίες των συναδέλφων στην συντριπτική τους πλειοψηφία διότι θέλω να έχουμε μια συλλογική δουλειά γιατί πιστεύω στη συλλογική δουλειά και όταν κανείς ε, συνεργάζεται με τους συναδέλφους του, βγάζει κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έκαναν τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σαλαβράκο. Ε, ξεκινάει λοιπόν η ψηφοφορία. Και έχουμε την τροπολογία υπερτιμών 21 του κυρίου Μάιερ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία η 48 του κυρίου Μάια, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 1, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 53 ε, της αδελφού Κολάσκα Μπομπίνσκα, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, μισό λεπτό ηλεκτρονικός έλεγχος, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ του αποτελέσματος. La Presidenza non è preparata. Anche la Vicepresidenza. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Eclipse psiforia. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ ψήφισαν και 7 ε, διαφώνησαν. Εγκρίνεται. Η 54 τη συναδέλφου Ζτανόκα, παρα, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, με συγχωρείτε, απορρίπτεται. Η 67 Κολάρσκα Μπομπίνσκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 55 καταπίπτει. Περνάμε στην 56 Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 του κυρίου Σαλαβράκου. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58, η 58 τροπολογία καταπίπτει η 59 του κυρίου Μπέκερ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Ζανόκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60, Κολάρσκα, Μπουμπίνσκα, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 62 Μάια υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε για την 62 του κυρίου Μάια. Έκλεισε η ψηφοφορία. απορρίφθηκε 15 υπέρ, ε, ναι, κατά. Κολάρσκα Μπομπίνσκα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 64 ε, Βαλέσσα ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 65 Μπαζέσκου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 66 Μπέκερ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται η 68 Κολάρσκα Μπομπίνσκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 70 του κυρίου Μάια υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 71 Στανόκα, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 17 του κυρίου Σαλαβράκου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 72 του κυρίου Μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 18 του κυρίου Σαλαβράκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 19 υπάρχει μια πρόταση προφορικής τροπολογίας ε, στην πρώτη πρόταση. Ε, διαφωνεί κανείς με αυτή την προφορική τροπολογία? Όχι. Κατόπιν τούτου ψηφίζουμε γιατί η 19 ως έχει τροποποιηθεί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 73 Μπαζέσκου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 74 Νέντελτσεβα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 Μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 76 αποσύρθηκε η 77 Καλόρσκα Μπομπίνσκα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 20 του κυρίου Σαλαβράκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αποσύρθηκε η 81, η 82 Σντανόκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 83 με ε, προφορική τροπολογία Διαφωνεί κανεί με την προφορική τροπολογία παρακαλώ. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 83 ως έχει τροποποιηθεί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 23 Κολάρσκα Μπομπίνσκα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 24 Κολάρσκα Μπομπίνσκα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 Μάια, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 26 υπέρ του κυρίου είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η παριθμόν 1 του κυρίου Σαλαβράκου υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2 του κυρίου Σαλαβράκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 του κυρίου Σαλαβράκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 4 του κυρίου Σαλαβράκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 27 του κυρίου Μάια υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 28 του κυρίου Μάγια υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 29 της κυρίας Βέρτμαν υπέρ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 30 του κυρίου Μάια υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 31 Μάια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 Μπέκερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 33 απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Λοιπόν, για την 33 του κυρίου Μπέκερ ψηφίζουμε. Non c'è dubbio che è stato approvato. 15 voti a favore, 8 contrari, l'emendamento... 15 υπέρ, 8 κατά, εγκρίνεται. Η 32 του Μάια υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 5 του κυρίου Σαλαβράκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 Μπαζέσκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 του κυρίου Σαλαβράκου υπέρ κατά κατά παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση, ε, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω από τα χέρια. Οι έξι ψηφίζουμε, του κυρίου Σαλαβράκου. Ψηφίζουμε παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε, έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία ε, 13 ε, κατά, 11 υπέρ. Η 7 του κ. Σαλαβράκου υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 35 του κ. Μάιερ υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 37 του κ. Μπέκερ υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 8 του κ. Σαλαβράκου υπέρ κατά, αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος, επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε για την τροπολογία υπερθμών 8 του κυρίου Σαλαβράκου. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Η τροπολογία απορρίπτεται. Η 36 Σντανόκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 38 Μπαζέσκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 του κυρίου Σαλαβράκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 του κυρίου Σαλαβράκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 39 Μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 40 μάια υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 44 η 45 του κυρίου Βαλένσα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 46 Μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 του κυρίου Σαλαβράκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 13 του κυρίου Σαλαβράκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 47 Μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 22 Κολάρσκα Μπομπίνσκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Eh, Ψηφίζουμε λοιπόν για το σύνολο του ψηφίσματος ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Άρχεται η τελική ψηφοφορία. 21 voti a 1 contrario. 21 υπέρ, 1 κατά. Συγχαρητήρια κύριε Σαλαβράκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που μας προσφέρατε και ευχαριστώ και όλους του υπόλοιπου συναδέλφους. Ε, τελειώνει, η, τελειώνει η ηλεκτρονική ψηφορία, μάλλον, η ψηφορία. Colleghi, vorrei riprendere i lavori. Ξαναξεκινάμε λοιπόν τις εργασίες μας. Ε, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες Επιτροπής Αναφορών για το 2011. Η συγητής είναι ο κύριος ο οποίος έχει και το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, μπαίνω στον πειρασμό να εκφράσω την ελπίδα ότι το γεγονός ότι η έκθεσή μου είναι στο σημείο 13 ε, της ημέρης διάταξης να μην είναι γρουσούζικο, να μην προϊονίζει κάτι κακό. Θα ήθελα να ακούσω και τους συναδέλφους να εκφράσουν τις απόψεις τους, αν έχουν βέβαια, για το τι πρέπει να συμπεριλάβει η εκθεσή μου, που νομίζω ότι θα είναι απλή, βασισμένη στα ε, γεγονότα στα πραγματικά στοιχεία για το τι έγινε πέρυσι, τι κάναμε στην Επιτροπή μας. Ούτως ή άλλως πρόκειται για την ε, πρώτη συζήτηση, έξω και περιμένω από τους αδέλφους ε, σχόλια και παρατηρήσεις για να τα συμπεριλάβω στο σχέδιο της εκθεσής μου. Όπως κατά το δυνατόν περισσότερες συστάσεις, ελπίζω να μπορέσω να συμπεριλάβω. Δεν θέλω να προδικάσω σε αυτή τη φάση το περιεχόμενο της έκθεσης. Ε, είμαι ανοιχτό να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων, άρα μπορώ να είμαι πολύ σύντομος. Ολοκληρώνω. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσίτσεστερ. Κυρία Άουκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ μια επιθυμία να είναι συγκεκριμένη η έκθεση. Το πλεονέκτημα της Επιτροπής είναι ότι εμείς έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ άλλες επιτροπές ασχολούνται πιο πολύ με αρχές. Εμείς ασχολούμαστε με συγκεκριμένες υποθέσεις. Γι' αυτό και κάνουμε και τις επισκέψεις αυτές τις διερευνητικές. Άρα δεν μιλάμε απλά, εργαζόμαστε κιόλας και αυτό θέλω να αντικατοπτρίζετε και στην έκθεσή σας. Αυτό είναι το βασικό μου αίτημα. Και βέβαια να αναφερθεί και η ακρόαση που είχαμε σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση. Βέβαια, ε, Κάποιες φορές αστάθηκα μήχανα γιατί για ώρα ήμουνα η μόνη που εκπροσωπούσα εκεί 500 εκατομμύρια κόσμο. Αλλά τέλος πάντων. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσίτσεστερ για την εισαγωγή που μας έκανε και για την πρόσκληση που μας απίφθινε να εκφράσουμε τις απόψεις μας για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών στη διάρκεια του έτους 2011. Ήταν και η πρώτη χρονιά που συμμετείχα εγώ ως μέλος στην Επιτροπή Αναφορών. 27 αναφορές από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία, τις πλέον πολυπληθείς χώρες της Ένωσης ε, κατατέθηκαν. Φυσιολογικό αυτό βέβαια. Είναι οι πολυπληθέστερες χώρες, άρα στατιστικά από αυτές τις χώρες παρέχονται και περισσότερες αναφορές. Είναι λογικό αυτό. Οι αναφορές οι οποίες αφορούσαν ε, οικονομικά θέματα ήταν πολυάριθμες και αυτό είναι φυσιολογικό λαμβανομένης υπόψης, υπόψη συγγνώμη, της οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ευρώπη. Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η συμπερίληψη του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην συνθήκη της Λισαβόνας και η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελούν ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες ε, μια δυνατότητα να μπορούν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους και για αυτούς τους τομείς. Οι πολίτες τείνουν να καταθέτουν αναφορές οι οποίες υπερβαίνουν το πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια καλή συνεργασία, μια αγαστή συνεργασία με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές για να μπορούμε να δίνουμε αποτελεσματικές απαντήσεις και να είμαστε αμερόληπτοι. Αυτό είναι ο στόχος μας. Ένα θέμα το οποίο συχνά συζητήθηκε μας απασχόλησε και στη πλαίσια της επισκέψης μας στη Ρουμανία. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω θα παραμείνει στην ιστορία των εργασιών της Επιτροπής μας. Να μιλάω για την ελευθεροτυπία. Ο κύριος Μποστινάρου γνωρίζω ότι έχει επιμείνει να αναδειχθεί το ζήτημα αυτό. Οι αναφορές για την ελευθεροτυπία κατά το έτος 2011 και αναφέρομαι συγκεκριμένα για τη Ρουμανία, ουσιαστικά ήταν μια ε, πολύ σημαντική για τη Ρουμανία, έξι για τη Βουλγαρία, για την Ουγγαρία επίσης, ήταν μια αναφορά και για την Ιταλία μια αναφορά. Άρα Μα νομίζω ότι η ελευθερία του τύπου είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται μόνο στη Ρουμανία και θεωρώ ότι το ζήτημα αυτό δεν θα πρέπει να το δούμε κομματικά. Όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας το κείμενο του κυρίου Τσίτσεστερ, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τη χρυσή τομή δεν θα πρέπει να γίνονται οι χώρες από την Ανατολική Ευρώπη ή από Πομπέι τράγοι. Θα πρέπει να έχουμε μια συνολική και ισορροπημένη εικόνα. Δεν θα ήθελα οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, επαναλαμβάνω, να γίνουν από δύο Πομπέι τράγοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εν γέννη η Ευρώπη. Θα είμαστε μάρτυρες φέτος και της πρώτης πρωτοβουλίας των πολιτών. Αλλά μάρτυρες και της ε, προσχώρησης ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θα συνταχθεί έκθεση και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε εξαιρετική συνεργασία και το 2012. Πρόεδρος, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Κύριε Τσίτσεστερ, έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ καθώς επίσης και τους συναδέλφους μου για τις παρεμβάσεις τους που με βοηθούν πολύ. Συμφωνώ με την κυρία Άουκεν ότι έχει σημασία η έκθεση να δείξει πόσο σκληρά εργάζεται η Επιτροπή Αναφορών, καθώς επίσης το βάθος και το εύρος των εργασιών της. Εμείς, τα μέλη της, είμαστε, θα έλεγα, μέλη μιας χρηστής λέσχης. Αλλά το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται στην παρούσα επιτροπή από την εμπειρία και σε άλλες επιτροπές και ιδίως αυτήν της βιομηχανίας όπου επίσης συμμετέχω ως μέλος ακόμη και αν το θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον δεν είναι πάντοτε εύκολο, εύκολο συγγνώμη, να παρακολουθούν τις ακροάσεις οι ε, βουλευτές. Ήδη τώρα γίνεται μία στην Επιτροπή Βιομηχανία και προφανώ δεν είμαι εκεί. Άρα συμβαίνουν τα πράγματα αυτά. Και σα κύριε Πρέντα, σα διαβεβαιώ ότι θα προσπαθήσω να επιτύχω μία ισορροπία. Είναι καθήκον και ευθύνη του εισηγητού αυτό και θα πράξω πάντο δυνατό για να την επιτύχω την ισορροπία αυτή. Θα εξετάσω προσεκτικά τα θέματα που θίξατε και θα τα περιλάβω στην έκθεση. Μετά την ανταλλαγή αυτή απόψεων θα προχωρήσω στην επεξεργασία του σχεδίου εκθέσεως που ελπίζω να ολοκληρώσω σύντομα και θα μπορέσουμε κατόπιν να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα επί της ουσίας. Κυρία Πρόεδρε, ή μάλλον κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εάν δεν έχετε να συζητήσετε τίποτε άλλο, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα, τότε πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίτσεστερ. Μπορούμε να περάσουμε, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, στο επόμενο σήμερα της μερικής διάταξης. Μετά από την ε, πρώτη Ανταλλαγή απόψεων λοιπόν για την Εθνική έκθεση για τη δραστηριότητα τη Επιτροπή Αναφορών. Περνάμε στο σημείο 14 αναφορά 13-27 2010 από τον Μωρίς Βίντς Γαλλικής Ιθαγένειας εξονόμητος των ενώσεων Αλζάς Νατίου και Ζεσεωνων Μεχσή η οποία συνοδεύεται από τρει υπογραφές σχετικά με το διάταγμα της Γαλλική κυβέρνησης τη 23 η Ιανουαρίου 2008 το οποίο χαρακτηρίζει τις εργασίες στη Μεγάλη Δυτική Παρακαμπτήρια Οδό του Στρασβούργου Α355 έργο κοινή ωφέλεια και επιγόντως απαραίτητες. Δεν ξέρω, είστε έτοιμος ε, κύριε να μιλήσετε. Θα περιμένουμε αν θέλετε, είστε έτοιμος. Όποτε θέλετε ξεκινάτε και καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε να συζητήσετε το θέμα το οποίο μας απασχολεί ε, και μάλιστα σπευσμένα μετά από την επιστολή που σας αποστήλαμε στις 27 Φεβρουαρίου. Περνά ο καιρό και είχαμε και μια ακρόαση 24 Μαΐου του 2011, όμως έκτοτε υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι σε πείσμα όλων και ενάντια σε όλους η Γαλλική Δημοκρατία θέλει να προχωρήσει αυτό το ε, σχέδιο. Ε, μετά, σε ό,τι αφορά μάλλον τη συγγραφή υποχρεώσεων, έχει θεσπίσει το κράτος τα κριτήρια της διαδικασίας επιλογής, ε, ε μικρή δημοσιονομική ε, δημόσια χρηματοδότηση, τεχνική ποιότητα, περιβαλλοντική ποιότητα, οικονομική ευρωστία και χαμηλά διόδια. Τελικά, ο Όμιλος Βίντσι, κατά μεγάλη μας έκπληξη, επελέγει, παρότι ήταν χειρότερη προσφορά του από όλα, σε όλα τα κριτήρια σε σχέση με τον ε, με τον όμιλο Ζάνεφ. Αν δείτε και το φάκελό μας 27 Φεβρουαρίου θα δείτε τα σχετικά στοιχεία. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι ε, η γαλλική δημοκρατία θέλει να δημιουργήσει τελικά προβλήματα, ιδίω ό,τι αφορά προστατευόμενα είδη όπω είναι το ευρωπαϊκό χάμστερ, ο πράσινο φρύνο και ο κοινό πυλοβάτη. Φαίνεται ότι ε, προτιμάει η κυβέρνηση τη Γαλλία να υποστεί τι οικονομικέ συνέπειε από την παραβίαση των ευρωπαϊκών οδηγιών και όχι να πει όχι σε αυτό το σχέδιο. 350 ε, εκτάρια ε, ζητά ο υποψήφιος και ε, τίποτα δεν έχει διαπραγματευτεί η κυβέρνηση για το χάμστερ, ενώ η Ζάνεφ ζητούσε 270 μόνο ε, εκτάρια. Και για το χάμστερ είχε κάνει κάποιες προτάσεις. Είναι ένα είδος πάρα πολύ ευάλωτο, προστατευόμενο. Εμείς γνωρίζουμε το έδαφος και μας δείχνει ότι οι αγρότες δεν πρόκειται να δεχθούν περαιτέρω προσπάθειες, ενώ ήδη τους επιβλήθη η επιλογή που έχει τις περισσότερες επιπτώσεις και μόνο η κατάληψη του σχεδίου ΖΕΣΕΟ θα μπορούσε να σώσει το χάμστερ αν ξανατεθούν δηλαδή από αμφισβήτηση αυτά τα 350 εκτάρια. Δεν καταλαβαίνουμε τους λόγους για τους οποίους κάνει ό,τι μπορεί η Γαλλική Δημοκρατία για να προχωρήσει αυτό το σχέδιο πριν τις επόμενες εκλογές και φαίνεται ότι δέχεται και τις συνέπειες που θα έχει, δηλαδή ότι τελικά θα εξαφανιστεί το αλζατικό, αλσατικό ευρωπαϊκό χάμστερ. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να σώσει το είδος αυτό και να, να προσπαθήσει να τηρηθούν οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Ε, θα δώσω τώρα στη συνάδελφό μου το λόγο για να μας πει για τα νομικά. Ε, δεν θέλω να επανέλθω στα επιχείρηματα που οποία σας έχουμε ήδη παρουσιάσει, αλλά θα ήθελα να επανέλθω ε, στην παραβίαση της οδηγίας 9243, ε, δηλαδή τη σχετική με τους οικοτόπους οδηγίας της 9 Ιουνίου του 2011. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε την ε, Γαλλία γιατί δεν τηρεί τις υποχρεώσεις ε, που ε, ενέχονται δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1 εδάφιο Δέλτα. Σας παρακαλούμε να μιλάτε λίγο πιο αργά. Je vais D'accord, pardon. Oui, d'accord, désolé. Donc voilà, donc c'était euh, des mesures, euh, c'était η απόφαση ε, αιτιολογήθηκε για το ότι δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα ε, για να πάψει η υποβάθμιση ή καταστροφή κάποιων χώρων αναπαραγωγής ή ανάπαυσης του ευρωπαϊκού ε, χάμστερ. Όμω με αυτό το σχέδιο βλέπουμε ότι υπάρχουν ελλείψει. Πρώτα απ' όλα το κράτο δεν έχει κάνει τίποτα για να προβλέψει αντισταθμιστικά μέτρα. Με βάση τα διακυβέρματα. τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία προτείνει το κράτο δεν επαρκούν. Το είχαμε ήδη πει τον Μάιο του 2011. Ενώ το κράτο δεν έλαβε και τα απαραίτητα μέτρα ώστε ήδη από τώρα να εξασφαλιστεί η δυνατότητα υλοποίηση των μέτρων αυτών. Η επιλογή του εργολάβου ε, γίνεται ενώ δεν περιλαμβάνει η προσφορά του κανένα ε, συγκεκριμένο αντισταθμιστικό μέτρο για αυτό το είδο Επομένω, Επομένως βλέπουμε ότι πολύ ελαφρά την καρδία αξιολογεί η Γαλλική Δημοκρατία την οδηγία για τους οικοτόπους. Δεύτερον, από την οδηγία που σα προανέφερα προκύπτει ότι υποβάθμιση και οι καταστροφέ θα είναι αναπόφευκτε για του χώρου παραγωγή και ανάπαυσης του ευρωπαϊκού χάμστερ δεν μπορεί να γίνουν παρά μόνο για επιτακτικούς λόγους μίζωνος δημόσιου συμφέροντος. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι αυτός ο αυτοκινητόδρομος δημιουργεί προβλήματα. Το 2005 είχε γίνει μια πυρογνωμοσύνη ανεξάρτητη από το ε, Γραφείο Μελετών ΤΕΤΕΚΑ της Καλσρούης που είχε δείξει ότι αυτό το σχέδιο που επελέγει και τις μεγαλύτερες επιπτώσεις θα έχει και τη λιγότερη αποτελεσματικότητα ε, θα είχε βλέπουμε ε, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θα δείτε με, τα, με τη σύγκριση αυτή που βλέπετε στη διαφάνεια, με τα μαύρα αυτά ε, σημεία. Ε, πρότεινε λοιπόν το TTK μια άλλη εναλλακτική λύση που θα σέβεται περισσότερο το περιβάλλον και θα λύνει και τα προβλήματα. Η τελευταία πρόταση. Η πρώτη όμω έχει επιλεγεί, που βλέπετε όμω ότι έχει και τρει κόκκινε κάρτες παρόλα αυτά. Ήδη λοιπόν τότε, αντί να έχουν συναρθεί επιπτώσει από αυτή τη μελέτη που είχε γίνει αποδεκτή, είχε, είχε χρηματοδοτηθεί, ε, τη θάβει αυτή τη μελέτη το, το κράτος. Άρα ε, πώς να δεχθούμε εμεί ότι υπάρχουν αυτοί οι τακτικοί λόγοι για το δημόσιο συμφέρον, αλλά αντίθετα ε, ε κατά την άποψή μου παραβιάζεται με το διάταγμα η Οδηγία 92 43. Δεν έχουμε χρόνο βέβαια να παρουσιάσουμε όλο τον προβληματισμό ε, για τη διάσωση του χάμστερ και τα άλλα περιβαλλοντικά ε, θέματα, αλλά γιατί η παράκαμψη αυτή προς τα δυτικά του Στρασβούργου θα βοηθήσει να διατηρηθεί το είδος αυτό που είναι βέβαια παρόν μόνο στην περιοχή μας. Πρώτα εξετάστε το τμήμα που είναι νότια του ΖΕΣΕΟ από το Piemont de Vos και που ξεκίνησε το 2009 το, το τμήμα αυτό και, και μπήκε σε κυκλοφορία από το 2011 φαίνεται εκεί με κόκκινο ότι παρόλα τα αντισταθμιστικά μέτρα και της διαπερατότητας του έργου δηλαδή με ειδικού αγωγούς για να περνούν τα χάμστερ αυτά βλέπετε ότι ο πληθυσμός του ζώου αυτού έχει ε, ε, αποχωρήσει εντελώς από εκεί. Και τώρα Βλέπετε ότι για την ώρα η διαπερατότητα αυτή δεν έχει παραμείνει παρά μόνο στα ευχολόγια. Η θέση του ΖΕΣΙΟ είναι λίγο διαφορετική. Αυτό πάλι είναι απλώς πιο μεγεθυμένη η ίδια διαφάνεια. Η κατάσταση του ΖΕΣΙΟ είναι λίγο διαφορετική, διότι οι πληθυσμοί που βρίσκονται στην περιοχή αυτή είναι πολύ λιγότερο πολυάριθμοι και δεν έχουν επαφή με τους άλλους πληθυσμούς, κάτι των ζώων αυτών δηλαδή, κάτι που είναι σημαντικό και για τη γενετική τους ανάπτυξη. Από όλους τους τομείς, εδώ αυτός ε, ο τομέας του πληθυσμού του ζώου αυτού έχει την περισσότερη την περισσότερη δυναμικό ανάπτυξης. Το έργο θα κόψει την περιοχή αυτή σε δύο, καθώς και τον πυρήνα του πληθυσμού, που δεν θα επιτρέψει επομένως την ανάπτυξη του χάμστερ. Είναι πολύ σημαντική η απόφαση που θα λάβετε για να μειωθεί η επίπτωση και να μην εξαφανιστεί το είδος αυτό από τη Γαλλία. Η γαλλική δημοκρατία δεν κάνει αρκετές προσπάθειες κατά τη γνώμη μας για να διασώσει το είδος αυτό. Το πέρασμα του αυτοκινήτου δρόμου αυτού θα είναι πια και η τελευταία πρόκληση και είναι καθαρή η διαφορία που δείχνει το κράτος για τη διάσωση του είδους. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους μας, να δώσουμε πρώτα το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, ε, κ. Ζωζέ Βαντεστέιεν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Οι αναφερόμενοι ανέπτυξαν την υπόθεση. Το διακύβευμα αναφέρεται στην διατήρηση τριών ειδών του μεγάλου χάμστερ, ενός και είδους βατραχιού και ενός άλλου είδους και η Γαλλία έχει καταδικαστεί ήδη από τον Ιούνιο του 2011 για την παράληψη λήψης μέτρων για τη διατήρηση των πληθυσμών του μεγάλου χάμστερ στην Αλσατία και αυτή είναι και η αιτιολόγηση. Κυρίως θεωρείται ότι παραβιάζεται το άρθρο 12 της οδηγίας περί που απαιτεί από τις χώρες μέλη να λαμβάνουν μέτρα για να διατηρηθούν τα είδη του παραρτήματος ε, της οδηγίας αυτής και σε αυτά περιλαμβάνονται το ευρωπαϊκό χάμστερο κοινό πυλοβάτης και ο πράσινος φρύνος που είναι τα τρία αυτά είδη που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ποια είναι η ανάλυση που κάνουμε εμείς τώρα της υποθέσεως. Μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Γαλλική Δημοκρατία υπέβαλε ορισμένε πληροφορίες την ενημέρωση των ε, μελετών επιπτώσεων επί του Ευρωπαϊκού Χάμστερ και των Βατραχιδών και αυτή έχει γίνει ήδη από το 2010 πρόκειται να λάβει μέτρα, ανεκκίνωσε, για να αποφευθούν οι επιπτώσεις ή να απαλληλθούν και να απαλληλθούν και οι παρελκόμενες επιπτώσεις με αντισταθμιστικά μέτρα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σημαντικό μέτρων. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε ε, πρόσθετες προφορίες, ιδίως για δύο θέματα. Πρώτον, για την αποτελεσματικότητα των συνιστομένων μέτρων. Θέλουμε δηλαδή διαβεβαιώσει σχετικά με την απετολισματικότητα των μέτρων που προτείνει να λάβει η Γαλλία και δεύτερον η Κομισιόν επιθυμεί να ε, ε, λάβει εγγυήσεις για την πραγματική λήψη των μέτρων. Όντω θα υλοποιηθούν τα μέτρα αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάληψη των ευθυνών του αναδόχου που έχει επιλεγεί θα ε, ελεγχθεί επίσης, θα εξεταστεί επίσης. Συνεχίζει την εξέταση του φακέλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το φως των πληροφοριών που έλαβε από τη Γαλλική Δημοκρατία για να δει εάν το έργο είναι συμβατό με την ανάγκη προστασίας των αναφερομένων ειδών. Ευχαριστώ κύριε Βαντεστέγεν. Οι ευρωβουλευτές τώρα έχουν το λόγο και πρώτα η κυρία Ρελιέρ Δεν θα επανέλθω στα γεγονότα τα οποία είχαμε ήδη συζητήσει προ λίγων μηνών και αναφερόμενοι τα υπενθύμησαν σήμερα. Η κατάσταση ε, έχει ως εξής. Υπάρχει η καταδίκη της Γαλλίας τον προηγούμενο Ιούνιο για ανεπάρκεια μέτρων που θα ήταν κατάλληλα να εξασφαλίσουν διατήρηση του είδους του ευρωπαϊκού χάμστερ. Η Κομισιόν σήμερα τόνισε και πάλι ότι εξακολουθεί να αναμένει ορισμένες πληροφορίες, πρόσθετες πληροφορίες δηλαδή για την αποτελεσματικότητα των προτινομένων μέτρων, για την αποτελεσματικότητα επίση των μέτρων που θα λάβει ο ανάδοχος. Από την άλλη μεριά, κανένα μέτρο μέχρι τώρα δεν έχει ληφθεί από την Γαλλική Δημοκρατία, από την καταδίκη και μετά, δηλαδή πάνω από ένα εξάμεινο, για την διαφύλαξη του είδους του ευρωπαϊκού χάμστερ. Και αυτό που είναι αρκετά εκπληκτικό συνεχίζονται οι ελιγμοί για να καταλήξουν σε ένα έργο δυτικά του Στρασβούργου και πρόκειται για ένα έργο το οποίο ήδη έχει αρχίσει να σχεδιάζεται εδώ και 50 χρόνια από τη δεκαετία του 1960 και διερωτάται κανείς και νομίζω νομίμως κατά πόσον είναι σχετικό πλέον το έργο αυτό διότι υπάρχει και μια σειρά μελετών που καταδεικνύουν ότι δεν πρόκειται να διευκολύνει τις αιχμές κυκλοφορίας την περιοχή του Στρασβούργου. 50 χρόνια χρειάστηκε να περάσουν δύο γενιές δηλαδή για να εξαλείψουν ένα είδος θηλαστικού από την γαλλική επικράτεια, το ευρωπαϊκό χάμστερ προκειμένου. Θα σας υποβάλω τη δική μου προσωπική ανάλυση, αλλά θεωρώ ότι προφανώς έχουμε εδώ ένα γαλλικό κράτος το οποίο έχει πεισματώσει να ε, συνεχίσει την, την υλοποίηση ενός προφανώς καταστροφικού έργου κατά παραβίαση των σχετικών οδηγιών χωρίς να λάβει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για τη διαφύλαξη ενός είδους θηλαστικού και αυτό που διαπιστώνει κανείς τους τελευταίους μήνες και ιδίω για την κατάσταση στη Γαλλία και την πολιτική κατάσταση λίγους μήνες μόλις πριν από τις προεδρικές εκλογές επιταχύνουν, αυτό φαίνεται καθαρά, επιταχύνουν την διαδικασία για να κλείσουν το θέμα αυτό, ώστε οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα της προεδρικής εκλογής, να μην μπορούμε πλέον να ανακρούσουμε πρίμνα. Η Γαλλία φαίνεται προτιμά να πληρώσει και να αναλάβει και τον κίνδυνο μιας νέας καταδίκης και επομένως και κυρώσεων, παρά να αναθεωρήσει ένα έργο που θεωρούν από ό,τι φαίνεται οι ασιατικές αλλά και οι γαλλικές αρχές ότι εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να μας πείσει ότι το έργο αυτό είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί. Διαρωτώ με εάν η Επιτροπή Αναφορών θα ήταν δυνατό να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει πίεση ώστε να παρασχεθούν και άλλες πληροφορίες και μάλιστα με επιταχυμένο τρόπο και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουλόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω ούτε εγώ να επανέλθω στο σύνολο του όλου προβλήματος για την παρακαμπτήρια αυτή οδό, δυτική οδό, δυτική αρτηρία. Η Γαλλία πράγματι καταδικάστηκε ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράληψη και αυτή η αρτήρια ουσιαστικά δεν φαίνεται να επιλύει το ζήτημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης ε, όπως θα έλπιζε κανείς. Λυπούμε επίσης, ε, όπως προϋπόθηκε, ότι τελικά φαίνεται ότι θα υπάρχει μεγάλη επίπτωση ε, στους οικοτόπους ε, όπου διαβεί το ευρωπαϊκό χάμστερ και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Παρ' όλα αυτά θέλω να μετριάσω λίγο ε, τα περί προεδρικών εκλογών που υπόθηκαν ή τέλο πάντων των βλεφτικών διότι όπως Είπαμε και όπως είπε και η προλαλήσα σας συνάδελφος, 50 ε, χρόνια υπάρχει αυτό το σχέδιο και έχουν γίνει και ξαναγίνει εκλογές. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα φορτώνουμε όλα στις πρόσφατες εκλογές, γιατί και παλιότερα θα μπορούσε να δοθεί έμφαση ε, για να μην ε, μπορούμε να γυρίσουμε πίσω κτλ. Ε, άρα μην δίνουμε πολιτική απόχρωση στο θέμα αυτό. Ελπίζω να μην χρειαστούν άλλα 50 χρόνια βέβαια, αλλά θεωρώ ότι για μια ακόμη φορά πρέπει να μην ενκτεί η συγκεκριμένη αναφορά, γιατί εκ νέου, γιατί ξαναβρισκόμαστε σήμερα, γιατί υπήρξαν νέα στοιχεία. Μας είπε πάλι η Κομισιόν ότι περιμένει ε, τεκμηριωμένη αιτιολόγηση από πλευρά Γαλλική Δημοκρατία για τα αντισταθμιστικά μέτρα. Άρα νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά εν αναμονή των απαντήσεων ε, που ελπίζουμε να είναι ακριβεί, σίγουρες και αποφασιστικές από την πλευρά της ε, Γαλλικής Δημοκρατίας για την ε, επιβίωση του είδους αυτού, του ευρωπαϊκού χάμστερ. Εγώ μπορώ να σας πω άκρος αντικειμενικά και χωρίς πολιτική απόχρωση ότι φαίνεται ενδιαφέρον αυτό το έργο, αλλά από την άλλη πλευρά αν υπάρχουν αποτελεσματικά αντισταθμιστικά μέτρα και αν αποδειχθεί ότι τουλάχιστον για το χάμστερ, γιατί μετά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την κυκλοφορία. Δηλαδή να έχουμε μια ε, μελέτη που να έχει κάποια αποτελέσματα. Τότε θα σκεφτούμε πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά νομίζω ότι θα μπορούμε πλέον να το εγκρίνουμε. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουλόν. Ακούσαμε τον κύριο Μπουλόν, δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προσθέσει κάτι. Να σας δώσω σε εσά ε, κυρίους και κυρία αναφέροντες. Έχετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα όσα είπε ο κύριος Μπουλό. Εμείς επίσης ε, λυπούμεθα που έχει πάρει και πολιτική διάσταση η συζήτηση αυτή αλλά με το έργο αυτό πραγματικά βλέπουμε ότι έχει επιταχυνθεί η όλη προσπάθεια. Δεν μπορούμε παρά να κάνουμε αυτή τη διαπίστωση. Δεν θα πάω πιο πέρα, αλλά τη διαπίστωση μπορούμε να την κάνουμε. Άκουσα τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την επιθυμία της για τα αντισταθμιστικά μέτρα και πράγματι πρέπει να δώσει απαντήσεις η Γαλλία και να είναι και αιτιολογημένες αυτές οι απαντήσεις. Γιατί Είμαστε στο, στη φάση της ολοκλήρωσης του δεύτερου σχεδίου δράσης ε, για το χάμστερ ε, και έχουμε και ένα τρίτο στάδιο. Είναι δυστυχώς αδύνατο να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Πάνω από 40 συνεδριάσεις είχαμε 1,5 μήνα τώρα. Όλα αυτά δείχνουν ότι ε, πολύ αραστεχνικά αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό. Εμείς καταλαβαίνουμε ε, ότι πρέπει να πατήσει η Γαλλία στην Κομισιόν. Δική μας όμως προτεραιότητα ακόμη και σήμερα είναι αποτελεσματικότητα, να μπορέσει να σωθεί αυτό το είδος. Το ευρωπαϊκό χάμστερ βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το είδος, έχουμε και την ε, αλσατική κοιλάδα με τη βιοπικιλότητά που πρέπει να διατηρήσουμε, όχι μόνο το χάμστερ. Ε, βλέπετε εδώ σε αυτή τη διάσταση, σε αυτή τη διαφάνεια ε, τις ε, μαύρες ζώνες, τις κόκκινες ε, και κάτω-κάτω βλέπετε τι μπορεί ακόμη να χτιστεί με τις κόκκινες ζώνες. Ε, βλέπετε τη σχέση, τη σύνδεση μεταξύ της νότια, του νότιου και του βόρειου πληθυσμού. Αν συνεχιστεί το έργο αυτό, θα αποκοπούν οι βόρειοι από τους πληθυσμούς. Θα δείτε λοιπόν να έχουμε τέτοια αποτελέσματα σαν αυτά που σας ε, δείχνω. Ε, θα, θα, θα σταματήσει να υπάρχει η συνέχεια. Ο πληθυσμός είναι πάρα πολύ ε, μικρός, 400 συγκεκριμένα είναι τα χάμσα τα οποία έχουν επιβιώσει και δεν ξέρω αν μπορεί πλέον να διατηρηθεί αυτό το είδος, τι δυνατότητες έχει όταν θα βλέπουμε να ε, εξαφανίζονται και άλλα εκτάρια γης. Ζητήσατε κυρία Μπουλόν να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Αν συμφωνείτε θα μείνει ανοιχτή και θα ζητηθούν από την ε, Γαλλία περισσότερες πληροφορίες. Και αφού ληφθούν αυτές τις πληροφορίες θα το ξανασυζητήσουμε. Συμφωνείτε? Ωραία. Ευχαριστώ. Μετά από το θέμα αυτό μπορούμε να περάσουμε στις ε, επόμενες αναφορές, αλλά αν με επιτρέπετε προηγουμένως ε, να πω κάτι που μου ζητάει γραμματεία να πω. Οι Ιρλανδικές είναι οι αναφορές που έπονται. Οι Ιρλανδοί συνάδελφοι είναι παρόντες, μάλλον θα έρθουν στις 10.30. Άρα μου ζητεί γραμματεία να κάνουμε έτσι μια διακοπή μέχρι τις 10.30 για να δούμε όλες τις αναφορές από κοινού. Το επαναλαμβάνω αφορούν ε, την Ιρλανδία όλες αν δεν διαφωνείτε συνάδελφοι, να κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 10.30 για να έχουν έρθει όλοι οι Ιρλανδοί συνάδελφοι και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Η κυρία Άουκεν βέβαια είναι εδώ. Ε, μόνο συμφωνείτε κυρία Άουκεν να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα και να συνεχίσουμε στις 10.30. Γιατί περιμένουμε τους Ιρλανδούς συναδέλφους. Λοιπόν, διάλειμμα μέχρι τις 10.30. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνονται οι εργασίες της Επιτροπής Αναφορών. Σας παρακαλώ κάνετε ησυχία. Επαναλαμβάνουμε τις εργασίες μας και περνούμε στο υπαριθμό 15. Είναι η αναφορά 161 του 2006, την οποία παρουσιάζει, έχει υποβάλει ο Νταν Μπρέναν, σχετικά με προβλήματα μόλυνσης στο Κιλκένι της Ιρλανδίας και τις επιπτώσεις στην τοπική κτηνοτροφία. Ο αναφερόμενος βρίσκεται στην αίθουσα. Έχετε τον λόγο κύριε Μπρέναν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σήμερα εδώ. Λέγομαι Dan Brenner ε, και έχω την ε, Jason, το αγρόκτημα. Ε, ο λόγος που κατέθεσα αυτήν την αναφορά είναι ότι δεν αναπτύσσονται σωστά τα βοηδή μας, τα ζώα μας. Είχαμε επιπτώσεις ε, στα ζώα μας. Ε, η δική μου, το δικό μου το αγρόκτημα εξετάστηκε από το Δεκέμβριο του 2002. Έχουν κατατεθεί πάρα πολλές αναφορές από τις Ιρλανδικές αρχές. Η τελευταία έκθεση που έγινε ήταν από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου και αυτό υπό τις εντολές του Υπουργείου Γεωργίας χρειάστηκε τρία χρόνια για να ολοκληρωθεί η μελέτη. Η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες αλλά δεν αναφέρονται οι παράγοντες αυτοί. Σε μια συνάντηση συνάντηση που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2012 με τους ερευνητές, μας είπαν οι ερευνητές ότι δεν γνωρίζουν ότι το Αμπονμπρίκ πλήττεται από το κάτμιο. Είπαν ότι δεν έχουν απάντηση για το τι συμβαίνει στο αγρόκτημά μας. Από τότε που έκλεισε το ε, εργοστάσιο ε, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε βέβαια κάποια βελτίωση. Στην συνάντηση διαπιστώθηκε ότι η έκθεση όμως που στάλει ε, από τις αρμόδιες αρχές ε, περιέχει πάρα πολλά κενά. Και δεν υπάρχει καμία απάντηση ε, γιατί για το κατά πόσο είναι σωστό ότι έκλεισε το εργοστάσιο και αυτό οδήγησε στο να υπάρξει σημαντική βελτίωση στην ανάπτυξη των ζώων στο δικό μου το αγρόκτημα. Alături de noi se află și reprezentanții ai Ministerului Agriculturii. Έχουμε εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας της Ιρλανδίας στην αίθουσα. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Μάτι Σέριντ. Ε, Madam Chairman. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας ε, για το ότι μας δίνετε την ευκαιρία στις Ιρλανδικές Αρχές να παρουσιάσουμε τη δική μας ε, την τοποθέτηση στις διάφορες εκθέσεις που εξετάζουν την περίπτωση. Είπα λοιπόν το όνομά μου και είμαι αναπληρωτής επικεφαλής ε, της κτηνιατρικής ε, μονάδας της υπηρεσίας μου. Έχω δεξιά μου τον αρμόδιο για την, ε, της υπηρεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ιρλανδία και επίσης και τον εκπρόσωπο από το Δουβλίνο και για της, ε, τον υπεύθυνο του, της μονάδας για ε, έρευνες, ε, επιδημιολογικές έρευνες, κυρίως για την περίοδο στην οποία αναφέρεται και η περίπτωση. Ετέθησα λοιπόν μια σειρά θεμάτων σε παλαιότερες συναντήσεις, κυρίως κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να απαντήσουμε σε αυτά που αναφέρονται στην επιστολή σας που στάλει το 2010 και εκεί γίνεται λόγος για την εφαρμογή της οδηγίας στην Ιρλανδία σε σχέση κυρίως με το εργοστάσιο Τούβλων. Η ε, Επιτροπή αναφέρει ότι διαπιστώθηκε μεγάλη περιεκτικότητα καδμίου στα ζώα. Ε, το αρμόδιο Υπουργείο για να έρθουμε εδώ, το αρμόδιο Υπουργείο και εμείς, ε, λέτε ότι Υπάρχουν προβλήματα στην κτηνοτροφική μονάδα του αναφέροντος ε, από το εργοστάσιο. Επίσης ε, γίνεται λόγος για το χρονικό διάστημα. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω μια έρευνα, ε, περίληψη των ερευνών που έγιναν για το θέμα του αναφέροντος και κατόπιν θα αναφερθώ στις εκπομπές Κατμίου. Ο κύριος ο αναφέρον έλαβε την άδεια λειτουργίας εξετάστηκε το θέμα του βάρους και της ενοχής. Ελπίζω λοιπόν ότι τα πορίσματα και τα συμπεράσματα που εξάγονται θα σας βοηθήσουν στο καθήκον σας να εξετάσετε αυτή τη συγκεκριμένη αναφορά. Να σας δώσω λιγάκι μια ιδέα για το πώς ακριβώς γίνονται οι έρευνες στην Ιρλανδία. Το πρόβλημα παραγωγής, όπως ε, λέει και αναφέρον, μας επισημάνθηκε στο τέλος του 2002 και αρχίσαμε να εξετάζουμε το θέμα το 2003. Έγιναν ε, έρευνες σε ζώα που είχαν πεθάνει και ε, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να διευρυνθεί η έρευνα για να εξεταστούν περιβαλλοντικοί παράγοντες συμπεριλαμβανομένης και της βιομηχανικής ρήπανσης. Υπάρχει ένα στάνταρ πρωτόκολλο που εμφαρμόστηκε το 2004 για να εξασφαλίσουμε το συντονισμό ανάμεσα στους διάφορους φορείς του κράτους που είναι αρμόδιοι για τέτοιου είδους έρευνες το Υπουργείο Γεωργίας και Αλίας και η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία αλλά και η αρμόδια υπηρεσία για την ασφάλεια των ε, τροφίμων. Αυτοί πήραν αναλύσεις από το έδαφος και από τα βότανα. Ε, Έγιναν αναλύσεις επίσης των εκπομπών από το εργοστάσιο ε, Τούβλων. Ενεπλάκη και υπηρεσία που είναι αρμόδια για την προστασία της υγείας ε, και τέλος ε, και η τοπική αρχή η οποία είναι αρμόδια για το πόσιμο νερό. Η ρημόδια αρχή στο Κίλκενι. Όλες λοιπόν οι έρευνες που έγιναν από το 2004 έγιναν υπό την καθοδήγηση της ομάδας, της διατομεακής ομάδας. Η τελική λοιπόν συλλογική έκθεση αυτής της διατομιακής ομάδας που αναφέρει τα πορίσματα των σοβαρών ερευνών που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 3 έως 9. Αυτά δημοσιεύτηκαν τον Αύγουστο του 2010. Σύντομα λοιπόν να πω το εξή. Σε αρκετές εκθέσεις και σε ένα έγγραφο που νομίζω θα σας βοηθήσει αναφέρονται τα πορίσματα αυτά. Ξέρω ότι δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο ε, και με μονομένε ε, εκθέσεις αναφορές ε, ε, μπορούν να έχουν και πάνω από 800 ε, σελίδες. Εγώ σας ε, προτείνω να διαβάσετε τις 12 σελίδες της περίληψης. Είδαμε λοιπόν τα πορίσματα όλων των αρμόδιων φορέων έρευνας και καταλήγουμε στο τελικό συμπέρασμα της διατομεακής αμάδας. Και σύμφωνα με αυτό το πόρισμα δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι προκαλείται ζημιά από τη βιομηχανική ρήπανση, ούτε ότι το κάδμιο προκάλεσε προβλήματα υγείας. Φαίνεται ότι υπάρχουν άλλοι πολλοί παράγοντες. Ε, θα μπορούσαν να έχουν προκύψει πολλές ε, ασθένειες ε, που οδήγησαν στην κατάσταση στην οποία περιγράφει ο αναφέρον και επίσης υπάρχουν και προβλήματα λήψεως αλάτων, όπως αναφέρεται. Διάφορες ερευνές αναφέρουν ότι είναι δύσκολο να γίνει εκτροφή στην περιοχή αυτή ε, όμως ε, η ποιότητα του εδάφους και των βοτάνων δεν είναι κακή. Η υπηρεσία της υγείας δεν εντόπισε ε, την αύξηση επικίνδυνων παραγόντων για την υγεία. Αυτή λοιπόν είναι η περίληψη της εργασίας που έγινε από τους κρατικούς φορείς στις επιστολές που σας ε, ανέφερα ε, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ότι πράγματι υπάρχει μεγάλη περιεκτικότητα καδμίου, ε, εντοπίστηκε αυτή στα ζώα. Το καδμίο αυτό μπορεί να αυξηθεί από τη βιομηχανική ρήπανση, να επηρεάσει τα ζώα, την υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Και το κάδμιο πράγματι μπορεί να προκαλέσει σημαντικά τοξικολογικά προβλήματα. Ε, πράγματι ε, στο αγρόκτημα του αναφέροντος εντοπίστηκαν μεγάλες περιεκτικότητες καδμίου, όμως δεν είναι αυτές ε, που προκάλεσαν το πρόβλημα. Η όλη ιστορία του καδμίου είναι πολύ περίπλοκη. Αρχικά λοιπόν είδαμε αύξηση του επίπεδου καδμίου στο αγρόκτημα, στους νεφρούς των ζώων. Επίσης πήραμε έκθεση από τον κύριο Κρίλι που είναι σήμερα εδώ παρόν σχετικά με τα επίπεδα καδμίου στο έδαφος και εκεί πράγματι ήταν αυξημένο το επίπεδο. Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος ε, κατέληξε ότι αυτό δεν είναι τόσο ανησυχητικό, διέταξε βέβαια περαιτέρω έρευνες και μας ζητήθηκε να το κάνουμε αυτό. Όλα αυτά έγιναν ως ε, ένα τμήμα των ερευνών που έλαβαν χώρα. Έγιναν, έγινε δείγματοληψία, ε, αίματος σε πάρα πολλά ζώα και εξετάστηκαν τα δείγματα αυτά για να διαπιστωθεί κατά πόσον ε, τα ζώα εκτέθηκαν σε κάδμιο ή σε άλλα βαρέα μέταλλα. Έγινε επίσης ανάλυση του εδάφους ε, στη επιτόπου. Αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ περίπλοκο και δεν έχει γίνει ποτέ στην Ιρλανδία. Ε, Τρεις νεφροί ε, ζώων μετά τη σφαγή τους εξετάστηκαν και υποβλήθηκαν σε περαιτέρω αναλύσεις. Τώρα, ως προς τις ε, αιματοληψίες, 3.000 περίπου αιματοληψίες έγιναν. Ε, υπήρξε ένα συγκεκριμένο δείγμα ε, και έγινε μια αρχική προεργασία πριν σταλούν τα δείγματα αυτά σε γερμανικό εργαστήριο. Και όταν ήρθαν πίσω διαπιστώθηκε ότι περίπου σε 600 ζώα διαπιστώθηκε ε, ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα καδμίου. Ε, στα άλλα 1.800 ή 1.700 περίπου δείγματα διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα καδμίου ήταν φυσιολογικά. Και όταν το εξετάσαμε αυτό κάναμε μία λεπτομερή εξέταση και διαπιστώθηκε ότι το εργαστήριο είχε κάνει λάθος. Είχε ε, κάνει ένα λάθος και υπάρχει μια πλήρης ε, έκθεση που εξηγεί ακριβώς τι συνέβη. Είναι στη μορφή παραρτήματος η έκθεση αυτή. Και τα δύο αποδεικτικά στοιχεία που θα σας αναφέρουν τα εξή. Υπήρχαν ε, ζώα ε, μακριά από το αγρόκτημα που παρουσίασαν τα ίδια αποτελέσματα. Όλα αυτά εμφανίστηκαν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή όταν επεξεργαζόταν το εργαστήριο τα δείγματα τα απόγευμα στις 2 η ώρα. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι το εμπορικό εργαστήριο, το ιδιωτικό εργαστήριο ε, που έκανε αυτό το λάθος, ε, το δέχτηκε, το παραδέχτηκε, είπε το λάθος είναι δικό τους. Έτσι λοιπόν, το μέρος εκείνο που φταίει, όταν το ομολογεί δηλαδή δημόσια το εργαστήριο και υπογράφει την έκθεση και λέει ότι έκαναν λάθος σχετικά ε, με το ότι αυτά τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα δεν είναι σημαντικά. Αυτό σας το έχουμε καταθέσει. Ένα άλλο θέμα είναι ε, τα επίπεδα background levels του καδμίου. Αυτό το συζητήσαμε με την υπηρεσία ε, που είναι αρμόδια για την προστασία των τροφίμων. Μας συνέστησε να συνεχίσουμε τις έρευνες και το κάναμε αυτό. Κάτι άλλο που κάναμε είναι το εξή. Οι δύο έρευνες που έγιναν για το έδαφος και για τα βότανα και δεν διαπιστώθηκε εναπόθεση καδμίου ε, στο έδαφος ή ε, στην υπόλοιπη βλάστηση. Άρα δηλαδή αν υπήρχε κάδμιο θα έφτανε στο έδαφος ή στη βλάστηση. Το τελευταίο θέμα που θέλω να πω για το κάδμιο είναι ότι πέρυσι κάναμε μία έρευνα για τα επίπεδα καδμίου ε, στα ζώα στην Ιρλανδία μετά από σύσταση της Επιτροπής Ασφάλειας Τροφίμων. Τα αποτελέσματα λοιπόν δείχνουν ότι τα επίπεδα καδμίου στους νεφρούς στα ζώα του κυρίου Μπρέναν δεν διαφέρουν ε, από το υπόλοιπο 25 μέχρι 30% ε, των ζώων στην Ιρλανδία. Υπάρχει κάποια μικρή αύξηση στα ε, background levels και τελικά ε, οδήγησαν αυτά στο υπάρχει μια συζήτηση για το κάτμιο στα ζώα. Το θέμα είναι ότι τα επίπεδα που διαπιστώθηκαν στα υπόλοιπα ζώα στην Ιρλανδία, 25 μέχρι 30%, ε, δεν διαφέρουν τα επίπεδα από αυτά που εντοπίστηκαν στην ε, μονάδα του κ. Μπρέναν. Άρα το κάδμιο δεν φταίει, μπορεί να φταίει οτιδήποτε άλλο. Και τώρα θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στον παρακαθήμενό μου, ο οποίος ε, θα αναλύσει το θέμα που έχει σχέση με το εργοστάσιο των τούβλων και εγώ θα επανέλθω για να ανακεφαλαιώσω. Ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω για την αδειοδότηση του τοπικού εργοστασίου παραγωγής ε, τούμπλων. Και τι επαφές είχαμε σε σχέση και με την διατομιακή αυτή έρευνα. Το EPA είναι ένα ανεξάρτητο φορέας που ιδρύθηκε το 1993 και έχει διάφορες ευθύνες, παρακολουθεί, αναφέρει, έχει σχέση με τις τοπικές αρχές, αναζητεί περιβαλλοντικές ευθύνες, συντονίζει την περιβαλλοντική έρευνα, προωθεί την ε, ε, τον περιορισμό των ε, θερμοκηπιακών αερίων κτλ. Το EPA έχει καθορίσει συγκεκριμένου κανόνες ό,τι αφορά την αδειοδότηση περιβάλλον, ε, μάλλον βιομηχανικών ε, δραστηριοτήτων και την επιβολή των κανόνων. Η εταιρεία η συγκεκριμένη συγκροτήθηκε το 68 ε, και πήρε το σημερινό της το 88 και παράγει τούβλα. Οι δραστηριότητες από το 99 και μετά μειώθηκαν και σταμάτησαν το Δεκέμβριο του 2008 εντελώς. Το EPA έδωσε, έδωσε άδεια το 2001 με βάση και τις καλύτερες δυνατές ε, τεχνικές. Δεν μεταφέρθηκε όμως η σχετική οδηγία την ε, εποχή της αδειοδότησης στο ελληνικό Δίκαιο, οπότε είχαμε μια τροποποίηση το 2006 για να ε, υπάρξουν διατάξεις ότι αφορά τη χρήση της ενέργειας, την πρόληψη των ατυχημάτων, και την παρακολούθηση κάποιων μεθόδων και για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Δόθηκε άδεια για τον έλεγχο των εκπομπών, για οριακές τιμές, για σχετικές παραμέτρους σε σχέση με τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στις διεργασίες. Οι οριακές αυτές τιμές για τις εκπομπές καθορίστηκαν για να μην υπάρχει περιβαλλοντική ρήπανση βασισμένη η διαδικασία αυτή στα, στα πρότυπα για την πέτα του αέρα και, για, και με χρησιμοποίηση μοντελοποίησης. Επίσης είχαμε κάποιες επιτόπου επισκέψεις και παρακολουθούσαμε τις τιμές ετησίως. Το Μάρτιο του 2003 ε, μας ενημέρωσαν για τα προβλήματα ε, στο αγρότημα του κυρίου Μπρέναν και εμείς λάβαμε μέρος σε αυτή τη διατομιακή έρευνα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Τροφίμων και εμείς ε, επικεντρώσαμε την έρευνά μας ε, στον ατμοσφαιρικό αέρα, την ποιότητα του αέρα συγκεκριμένα, για το ενδεχόμενο ρήπανσης ε, και ειζημάτων, αναπόθεσης καδμίου. φθόριο βρήκαμε ότι απελευθερώνεται κατά τη ε, διαργασία κατασκευής των ε, τούβλων. Οι εκπομπές από το εργοστάσιο, τα αρχεία παραγωγής, εκτίμηση των πρώτων υλών ε, και η μοντελοποίηση παρακολουθήσαμε τα επιφανειακά, τα υπόγεια ύδατα, τις, ε, τα βαρέα μέταλλα, ε, το πεχά και άλλα. Σε ό,τι αφορά το κάδμιο, αναλύσαμε τις πρώτες ύλε και είδαμε πολύ χαμηλή υπερεκτικότητα ε, καδμίου και πολύ ελάχιστες απώλειες, έκκληση καδμίου στην ατμόσφαιρα. Το 2004 και το 2005 δεν εξήχθησαν οι σχετικές έρευνες. Το 2004 δεν είχαμε σύμπτωση για των αποτελεσμάτων ε, για τα 0,5 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο. Ούτε είχαμε το 2005 ενδείξεις για έκκληση καδμίου σε σημαντικά επίπεδα. Το EPA έκανε και μοντελοποίηση για την διάχυση καδμίου, διασπορά καδμίου και την εναπόθεσή του στην ε, τέφρα, στην σκόνη και ούτε και εκεί είδαμε να υπάρχουν ε, εκπομπές καδμίου από αυτό το εργοστάσιο. Και βασιστήκαμε σε κάποια δεδομένα τα είχαμε λάβει από τις αρχές του 2004 σε ό,τι αφορά την ανάλυση του εδάφους ε, και του ε, γρασιδιού έδειξαν ότι δεν υπάρχει ούτε και εκεί αναπόθεση κατά σε σημαντικά επίπεδα. Το EPA λοιπόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπομπές ε, καδμίου είναι περιορισμένες από το εργοστάσιο, δεν έχουν οδηγήσει σε σημαντική περιβαλλοντική ε, επίπτωση. Το 2007 Προσλάβαμε διεθνούς, ε, διεθνείς εμπειρογνώμονες ε, και από την περιβαλλοντική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και κάποιους από τις ΗΠΑ, οι οποίοι έκαναν μία αξιολόγηση από νοτήμους ε, και είδαν και το κατά πόσον τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία. Έκαναν επιτόπιες επισκέψεις στο εργοστάσιο, παραγωγής τούβλων, μελέτησαν τα αρχεία αδειοδότησης κτλ. Και κατέληξαν στο ότι ε, είχε γίνει η έρευνα από το EPA με βάση τις βέλτιστες δυνατές ε, πρακτικές και τεχνικές. και ότι είχαμε κάνει ό,τι μπορούσαμε για να ελαχιστοποιήσουμε τις εκπομπές από αυτό το εργοστάσιο. Στην διατομιακή έκθεση συνοψίζονται τα πορίσματα της ε, υπηρεσίας μας. Και όπως σας είπα, Εκεί περιλαμβάνεται μια εκτεταμένη ανάλυση που δείχνει ότι δεν βρήκαμε ότι υπάρχει ε, κλίση κάποιων ε, επιβλαβών ουσιών. Και δεν υπάρχει απόδειξη ότι είτε το φθόριο είτε το κάδμιο ευθύνονται για τα προβλήματα στο αγρόκτημα του κύριου Μπρένα. Uh, Δύο θέματα κυρία Πρόεδρε. Πρώτο, η προσέγγιση για την αξιολόγηση των, των ε, δεδομένων, των ενδείξεων και δεύτερον για την αντίληψη των αιτίων που οδήγησαν στο πρόβλημα. Και αναφέρομαι στην έκθεση 2009 που περιλάμβανε κάποια βασική έρευνα αλλά κυρίως την συλλογή και αξιολόγηση όλων των υφισταμένων δεδομένων. Εξετάσαμε 15 μελέτες που ήταν διαθέσιμες ορισμένες που είχαμε κάνει εμείς άλλες από την Ιρλανδική κυβέρνηση και ορισμένες ανεξάρτητες και 7 ε, αναλύσεις υποστήριξης που κάναμε. Το βασικό ερώτημα που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε ήταν υπήρχαν ενδείξεις που να στηρίζουν κάποια από τις ακόλουθες υποθέσεις ειδική για την ε, διαχείριση της, ε, του αγροκτήματος τη γενετική, την διατροφή των ζώων κλπ. και άλλες υποθέσεις που δεν ήταν συγκεκριμένες, δηλαδή για περιβαλλοντική μόλυνση, άλλες ελλείψεις κλπ. Και το αποτέλεσμα ήταν ε, η συγκεκριμένη υπόθεση μπορούσε να εξηγήσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Νταν Μπρέναν. Κάθε μια από τις υποθέσεις και όλα τα σχετικά δεδομένα που είχαν σχέση με την κάθε μια υπόθεση αξιολογήθηκαν με αντιπαραβολή με τα γνωστά διεθνή κριτήρια κριτήρια τα οποία είναι κατάλληλα για να επιτρέψουν σε κάποιον να κατανοήσει και να θέσει σε δοκιμασία και να εξετάσει εάν υπάρχει ε, κάποια σχέση συνάφειας μεταξύ των ενδείξεων και της υποθέσεως. Το άλλο που είναι σημαντικό νομίζω για την ε, Επιτροπή σας είναι ότι όσο οι υποθέσεις γίνονται πιο περίπλοκες και τα δεδομένα είναι περισσότερα, είναι επόμενο να υπάρχει κάποια αβεβαιότητα σχετικά με τα συμπεράσματα διότι ορισμένα δεδομένα στηρίζουν κάποιε από τις υποθέσεις αυτές και άλλα όχι. Εν ώψη λοιπόν αυτή της αβεβαιότητας η προσέγγιση που επιλέξαμε και που είναι ανάλογη με αυτήν που γίνεται για παράδειγμα και για την αλλαγή του κλίματος αλλά και άλλα παρόμοια όπου υπάρχει δηλαδή ένα στοιχείο αβεβαιότητας είναι να εξετάσουμε τις ενδείξεις και, το βάρος της αποδείξεως με μια κλίμακα από 0 έως 10. Δηλαδή 0 ουδεμία απολύτως ένδειξη μέχρι το 10 που σημαίνει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία ότι η υπόθεση, η συγκεκριμένη υπόθεση δηλαδή που κάνουμε είναι αληθής. Το 5 θα ήταν το αντίστοιχο με μια υπόθεση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, ενώ το 9 θα ήταν η απόδειξη που απαιτεί ένα ποινικό δικαστήριο, δηλαδή πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας. Εμείς φτάσαμε στο 5 αντίστοιχο δηλαδή με μια αστική δίκη που θα κάνει μια ε, αξιολόγηση των πιθανότητων. Αυτή είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποίησαμε. Το ενδεχόμενο τώρα το εργοστάσιο να είναι η αιτία ή να έχει συμβάλει αρνητικά εννοείται στην αρνητική απόδοση των γελαδιών του Ουντάν, εμείς είχαμε πληροφορίες κυρίως από 10 διαφορετικές πηγές. Η να εχει συμβαλει αρνητικα εννοειται στην αρνητικη αποδοση των γελαδιων του Νταν. εμεις ειχαμε πληροφοριες κυριως απο 10 διαφορετικες πηγες η πρωτη έχει σχέση με τα γεγονότα και πότε αυτά συνέβησαν, πότε άνοιξε το εργοστάσιο, πότε έκλεισε το εργοστάσιο. Τέσσερι ήταν οι γενικέ μελέτε, ορισμένε που έγιναν από την υπηρεσία μα EPA, άλλοι από, άλλες μάλλον από ανεξάρτητους επιστήμονες, δύο μελέτες ειδικά για το φθόριο και μία για το κάδμιο. Με όλε αυτέ τι υποθέσει ξεκινήσαμε πάντοτε από το βαθμολόγιο 0, δηλαδή να μην υπάρχει πολύ καμία ένδειξη υπέρ της υποθέσεως και μετά εξετάσαμε όλες τις ενδείξεις. Και σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να τα προκαλεί αυτά το εργοστάσιο, φτάσαμε περίπου στο 2 3. Με την έννοια ότι το 2 είναι πιθανόν, το 3 είναι εύλογο και στηρίζεται από ορισμένε ενδείξεις. Αυτά με βάση τα δεδομένα που είχαμε στη διάθεσή μας στα μέσα του 2009. Δηλαδή ασθενείς μόνο ενδείξεις υπάρχουν υπέρ της υποθέσεως ότι ευθύνεται το εργοστάσιο. Και μακριά είναι και από το 5 που θεωρήσαμε, όπως είπα προηγουμένως, ότι είναι το κατόφλι που ε, κάναμε την αντιπαραβολή. Στις περισσότερες από τις 10 μελέτες δεν υπήρχαν καν ενδείξεις υπέρ της υποθέσεως του εργοστασίου. Έρχομαι τώρα στην ερμηνεία μας των δεδομένων σχετικά με την περίοδο όπου το ε, εργοστάσιο άνοιξε και μετά έκλεισε και σας υπενθυμίζω ότι το έργο μας έχει σχέση γίνει ότι περίπου τα μέσα του 2009. Από το 2003 έως το 2008 που διήρκεσε η μελέτη μας, το εργοστάσιο έκλεισε για δύο σχετικά μικρά χρονικά διαστήματα, αρχές του 2007 και αρχές του 2008. Σε αυτές τις περιόδους κλεισίματος του εργοστασίου ήταν καλή η απόδοση των γελαδιών, αλλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι το, η καλή ήταν απόδοση των ζώων και σε ορισμένε άλλε περιόδους όπου το εργοστάσιο ήταν ανοιχτό. Βασισμένη λοιπόν με βάση μόνο αυτές τις ενδείξει, δεν μπορεί κανείς να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για το αν το εργοστάσιο συνέβαλε στο πρόβλημα. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι ήταν σημαντικό να μετρηθεί η απόδοση των ζώων όταν έκλεισε το εργοστάσιο του 2008 και το προσωπικό μου προσφέραμε την υποστήριξή μας στον Ντάν για να το κάνουμε αυτό, αλλά την απέρριψε επιμόνως. Τα δεδομένα των τελευταίων ετών, ωστόσο, δείχνουν μια σημαντική βελτίωση της απόδοσης σε γάλα των ζώων. Μέχρι τώρα δεν έχουμε όμως συγκεκριμένα δεδομένα, εκτός από την απόδοση των Μοσχαριών το 2009, δηλαδή τη χρονιά μετά που έκλεισε το εργοστάσιο. Εκείνη τη χρονιά δεν υπήρξε ωστόσο καμία αντικειμενική βελτίωση που να παρατηρήθηκε. Δεν μπορώ να σχολιάσω ε, δεδομένα των 2010 έως 2012 ε, γιατί δεν έχω τέτοια. Τώρα, τα δεδομένα σχετικά με την περίοδο που ήταν ανοιχτό το εργοστάσιο και πότε έκλεινε, αν ήταν θετικά, θα ήταν απίθανο από μόνα τους να μεταθέσουν το βάρος αποδείξεως από το κατόφλι του 5 και πάνω. Θα χρειαζόντουσαν λοιπόν και άλλες ενδείξεις. Αυτή η περίοδος, οι χρονικές περίοδοι δηλαδή του κλεισίματος και του ανοίγματος του εργαστασίου πρέπει να ελεγχθούν και με βάση άλλες παραμέτρους που άλλαξαν μέσα σε αυτή την ε, περίοδο των 10-15 ετών. Ευχαριστώ θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, <clears throat> ένα λεπτό μου επιτρέπετε ακόμα. Ακούσατε σημαντικές διαφορές απόψεων ως προς την ερμηνεία των πορισμάτων των εκθέσεων ε, της ε, διατομιακής ομάδας. Στην πρόσκλησή σας αναφέρεται ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το εργοστάσιο τούβλων προκάλεσε το πρόβλημα. Εμείς λέμε σήμερα ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για να στηριχθεί αυτή η άποψη. Πάντως, αυτό που μπορεί να γίνει στην προσπάθειά σας ως ουδέτεροι παρατηρητές ε, είναι τις εκθέσεις αυτές ε, να τις παραπέμψετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσετε να παραπεμφθούν από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ σε ένα κοινό ερευνητικό συμβούλιο ή στην ΕΨΑ. Ε, οι Ιρλανδικές αρχές και οι συντάκτες της έκθεσης ε, με μεγάλη τους χαρά να μιλήσουν λεπτομερώς για το θέμα αυτό με τους εμπειρογνώμονες ε, και η Επιτροπή Αναφορών θα μπορούσε να έχει και αυτή έναν δικό της άνθρωπο για να καταλήξει στα συμπεράσματά του. Και μου επιτρέπετε να σας προτείνω αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Um, um, Σας ευχαριστώ. Λίγα λόγια για τα θέματα που έφυξε το Υπουργείο. Δεν νομίζω ότι η υπηρεσία EPA ήταν ιδιαίτερα διαφανής σε ό,τι αφορά την καταγραφή των ε, εκπομπών ρήπων καδμίου από το εργοστάσιο. Κάτι άκουσα, δεν κατάλαβα πολύ καλά. Η πραγματικότητα είναι ότι τον Απρίλιο του 2004 η υπηρεσία EPA βρίσκει 24 γραμμάρια την ώρα. Δηλαδή 160 φορές παραπάνω από τις ε, κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν και για το κάδμιο. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι 0,5 γραμμάρια, ενώ σύμφωνα με την Κομισιόν 24. Ίσως να τα ακούσατε αυτά από, ίσως να τα ακούσατε αυτά από την EPA, εγώ δεν τα άκουσα. Όταν λοιπόν συμπεραίνουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εκπομπές καδμίου από το εργοστάσιο μπορεί να έχουν ε, προκαλέσει τα προβλήματα στα γελάδια του Νταν, αυτό δεν είναι αλήθεια. Και 200 δείγματα αίματος ήταν μολυσμένα από το αγρόκτημα αυτό και αυτά ελέγχθηκαν σε εργαστήριο εγκεκριμένο από την EPA. Ήδη όμως πριν είχαν βρεθεί δείγματα αίματος από τα ζώα με 200 μιλιγράμμ και πάνω, 1000 γραμμάρια και πάνω. Τοξικά για τον άνθρωπο. Πριν από, πριν από αυτήν την ε, ρήπανση βρήκανε 200 μιλιγράμμ. Και μετά από λίγους μήνες βρήκαν μάλιστα ένα, σε ένα ζώο 400 μιλιγράμμ καρμίου νομίζω ότι δεν προέκυψαν σαφώς αυτά από την κατάθεση των μελών του Υπουργείου. Βρήκαν πιθανώς τοξικά επίπεδα καδμίου στο αίμα των γελαδιών του Ντάν, ανεξαρτήτως από το που προέκυψε αυτή η ρήπανση. Πώς είναι δυνατόν να μολύνθηκαν σε εγκεκριμένο εργαστήριο με καθαρό κάδμιο. Δεν υπάρχει το κάδμιο αυτό πάνω στα τραπέζια του εργαστηρίου για να πήγε να μολυνθεί το αίμα από εκεί, όμως συνέβη και όταν αυτοί είχαν το αίμα στην διάθεσή τους. Και ένας αριθμός δειγμάτων εξαφανίστηκαν. Οι ερευνητές έλαβαν δείγματα δύο μήνες αργότερα, δεν τα εξέτασαν ποτέ διότι τα έχασαν. Όλα τα δείγματα από, την, από το αγρόκτημα του Ντάν χάθηκαν. Η Κομισιόν θα σας πει ότι το εργοστάσιο είχε συμμορφωθεί στην ε, νομοθεσία. Έκαναν μια ανεξάρτητη εκτίμηση και ότι έκαναν καλή δουλειά για να μειώσουν τις εκπομπές. Αλλά το έργο αυτό έγινε με έναν online fluoride ε, ε, counter, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο παρακολουθεί τις εκπομπές φθοριούχου άλατος online, επιγραμμικά. Είπαν, είπε η ίδια η Επιτροπή όμως ότι θέλει να εξετάσει ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας τον μετρητή αυτό και αποδείχθηκε ότι έκανε λάθος μετρήσεις. Αντί 21 που λάμβανε μετρούσε 10 μονάδες. Και αυτό νομίζω επίσης δεν ακούστηκε από τους εμπειρογνώμονες του Υπουργείου. η Προεδρεύουσα. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο στο τέλος της συζητήσεως. Θα δώσω το λόγο στον δεύτερο ε, αναφερόμενο. Να επανέλθω κι εγώ στον Μάικλ Σέρτον που πολύ σωστά είπε ότι υπήρχαν τέσσερα συμπεράσματα, τέσσερα πορίσματα ε, στην διατομιακή έρευνα. Χαίρομαι γιατί ανέφερε την έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στο Index Farm ε, ήταν ε, δύσκολο ε, να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα ότι σε πολλά αγροκτήματα το έδαφος και τα βότανα μοιάζουν, αλλά δεν μας είπε ότι δεν ήταν οι ίδιες οι πρακτικές σε αυτό το αγροκτήμα σε σχέση με άλλα αγροκτήματα, ότι δηλαδή δεν ήταν υπεύθυνε πρακτικές που ε, ασκεί στο ε, αγροκτημά του ο Νταν Μπρέναν. Επίσης είπε ότι δεν υπήρξαν κάποια συνήθη πρότυπα ή κάποιες ανθρώπινε γνώσει στην περιοχή, αλλά ποτέ η καποιες ανθρωπινες γνωσεις στην περιοχη αλλα ποτε η αρμόδιοι δεν ήρθαν στο αγρόκτημα, δεν μίλησαν ποτέ με μέλη της οικογένειάς τους, ούτε πήραν ποτέ τα ιατρικά τους αρχεία. Υπάρχει κάποιος άλλος ε, από τους αναφέρους που θα θέλει να λάβει το λόγο, αν όχι να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής... Η Πρόεδρος για δεύτερη φορά με διακόπτεται, Θα δώσουμε το λόγο πρώτα στην Κομισιόν. Θα έχετε εσείς μετά το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω λίγο για την έρευνα την οποία έχει ξεκινήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτό το εργοστάσιο πληθοποίησης και τις αποδόσεις, τις επιδόσεις του σε σχέση ε, με την οδηγία την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο του, την οδηγία του 96. Είναι μια οδηγία που την ε, λέμε στον τομέα IPPC και απαιτεί εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν ε, στο πεδίο εφαρμογή της να εφαρμόζουν ε, τις καλύτερες δυνατές τεχνικές για την πρόληψη και την ελεγχιστοποίηση των εκπομπών. Και η οδηγία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, μεταξύ αυτών και η κεραμοποιία και στην προκειμένη περίπτωση το πληθοποιείο το συγκεκριμένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έλθει στην Επιτροπή σας κάποιες φορές για να συζητήσει τα πορίσματά της και προσπαθούμε να συνοψίσουμε τα πορίσματα και των δικών μας επισκέψεων αλλά και σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για τις άδειε και για την παρακολούθηση, τα στοιχεία που λάβαμε. Θα τα σχολιάσω. Η πρώτη σύγκριση έχει να κάνει βέβαια αφενός ε, με τους όρους αδειοδότησης ε, του εργοστασίου κατασκευής πλήνθων και αυτό το οποίο εμείς συνιστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, ως ισοδύναμη τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές. Και για το στόχο αυτό έχουμε ένα έγγραφο αναφοράς Μπρεφ λέγεται αυτό, για τι βέλτιστες δυνατέ τεχνικέ. Αυτό περιλαμβάνει τι τυπικέ εκπομπέ που αναμένει κανεί ε, με την εφαρμογή των καλύτερων δυνατών τεχνικών. Πρώτη σύγκριση λοιπόν ήταν μεταξύ αυτού του εγγράφου αναφοράς ε, BAT και των στοιχείων που έχουμε. Και βλέπουμε ότι οι άδειε εν γέννη εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο του BAT. Και σας το έχουμε πει και σε προηγούμενη επίσκεψη μας στην Επιτροπή σας. Η επόμενη έρευνα που κάναμε βασίστηκε στα στοιχεία παρακολούθησης ελέγχου. Στη, συγκρίναμε τα στοιχεία ελέγχου με τις, προϋποθέσεις για την ε, έγκριση της άδεια. Και τι είδαμε στην πιο πρόσφατη έρευνα που διεξαγάγαμε. Είδαμε ότι μεταξύ της περίοδου 2001 και 2006 υπήρξαν κάποιες παραβιάσεις ε, των όρων αδειοδότησης οι οποίες σχετίζονταν κυρίως ε, με τις εκπομπές φθορίου και σε δέκα περιπτώσεις το είδαμε αυτό, για χλωριού χάλατα ορισμένες φορές και για το τα οξύδια ζώτου μία φορά. Η... Τα στοιχεία τα οποία συνέλεξαν οι Ιρλανδικές αρχές περιλαμβάνουν κάποιες διορθωτικές δράσεις για το εργοστάσιο κατασκευής πλήνθων για να διορθωθούν αυτές οι παραβιάσεις. Τώρα, αφού είδαμε το, την άδεια. Είδαμε την μη συμμόρφωση και τι δράσεις ανέλαβαν οι Ιρλανδικές αρχές. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε εμείς ε, να προσδιορίσουμε μέσα στην οδηγία IPPC για την άδεια είναι παραβία της οδηγίας της συγκεκριμένης. Οι πληροφορίες που έχουμε εξετάσει είναι 2001-2006, τα στοιχεία 2001-2006. Οπότε με βάση τις πληροφορίες τις οποίες εμείς αξιολογήσαμε που είχαμε λάβει η μη συμμόρφωση είναι αυτό που σας εξέθεσα. Κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι οδηγιά η PPC ετέθη πλήρω σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Οκτωβρίου 2007. Και μένω σε αυτά. Ευχαριστώ. În continuare voi da cuvântul doamnei Prendergast. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε ε, λύση. Αυτό είναι προφανέ σε όλου μα. Υπήρξε επίση μεγάλη σύγχυση σε σχέση και με τα, τα επιστημονικά στοιχεία τι διάφορε εκθέσει, οι οποίε έχουν αναφερθεί από τι διάφορε Ιρλανδικέ αρχέ. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν κυρία Πρόεδρε να παραπέμψετε και την ε, αναφορά και τα επιστημονικά στοιχεία και τις εκθέσεις ε, ε, στο Γενικό Συμβούλιο για να γίνει μία ανάλυση. Διότι αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο εμείς ως βουλευτές να καταλήξουμε σε λογικά ε, συμπεράσματα σε σχέση με το τι θα πρέπει να κάνουμε με αυτήν την ε, αναφορά. Θα την αρχιοθετήσουμε ή όχι. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες. Όπως ξέρετε δεν είμαι πια μέλος αυτής της Επιτροπής, αλλά ήμουν μέλος όταν ήρθε για πρώτη φορά εδώ ο κύριος Μπρέναν. Και είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι αυτή η αναφορά υπάρχει στην Επιτροπή μας ε, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση. Εμείς ε, νιώθουμε συμπάθεια για το πρόβλημα του κ. Μπρέναν και θέλουμε να τον στηρίξουμε να βρεθεί κάποια λύση. Παρά τα αρνητικά στοιχεία υπάρχουν και δύο θετικά που προέκυψαν σήμερα το πρωί. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι για πρώτη φορά νομίζω έχουμε εκπροσώπους από κράτος μέλος οι οποίοι εκπρόσωποι ε, επιθυμούν να ενημερώσουν σχετικά με μια συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό είναι πολύ καλό και είναι και ευχάριστο επίσης το να ακούμε ότι η κατάσταση ε, στο αγρόκτημα βελτιώθηκε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπα την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, δηλαδή ότι πράγματι χρειαζόμαστε για το θέμα αυτό επιστημονική παρέμβαση. Γιατί ακούει κανείς από τις δύο πλευρές ότι δεν συμφωνούν ακόμα και για κάποια ε, συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν επιστημονικές εκθέσεις στην Ιρλανδία. Ε, διαφωνούν κάθετα ως ε, προς τις εκπομπές που περιέχουν κάδμιο και γι' αυτό λοιπόν νομίζω θα ήταν χρήσιμο η Επιτροπή να κάνει αυτό που είπε ο κ. Σέραντον, δηλαδή να ε, παραπεμφθεί η Επιτροπή σε κάποιο αρμόδιο φορέα, έτσι ώστε η Επιτροπή να μπορεί να έχει μια γενική εικόνα των αποδεικτικών στοιχείων και να μπορεί μετά να δώσει την κατεύθυνση. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή να σχολιάσει αυτή την πρόταση, αν θέλετε, δική μου και να μας πει επίσης και ο κύριος Μπράναν ο ίδιος τι πιστεύει για την πρόταση αυτή, ε, γιατί θέλω να μας πει αν στηρίζει αυτή την άποψη. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η δική του η άποψη, γιατί η Επιτροπή αυτή τη τελική ανάλυση έχει στο επίκεντρο τον πολίτη. Αν λοιπόν ο αναφέρον είναι ανοιχτός σε αυτή την πρόταση και αν τα κρατημέλη επίση είναι πρόθυμα να δώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να συνεργαστούν και αν υπάρχουν και αρμόδιοι φορείς να γίνει η σωστή δουλειά, νομίζω αυτός είναι ο καλύτερος για για να ε, ολοκληρωθεί η υπόθεση. Γιατί όλοι μας γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι υπήρχε πρόβλημα. Το να λέει κανείς ότι τα αίτια είναι πολλαπλά, ίσως να είναι. Αλλά αυτό δεν ε, ικανοποιεί τον αναφέροντα και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Ίσως ε, να μας πει η Επιτροπή την άποψή της αυτό που είπα, αλλά και ο αναφέρον να μας πει και αυτός, να μας πει κατά πόσο στηρίζει αυτή την πρόταση και υπό ποιες προϋποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό ενδιαφέρον για την υπόθεση γιατί είναι εκτός της εκλογικής μου περιφέρειας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο αναφέρον. Μπαίνω στη θέση του λοιπόν. Και πρέπει να πω ότι είναι καλό που ακούμε σήμερα ε, και τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν συμμετείχε και παλαιότερα το κράτος σε αυτή την υπόθεση. Ίσως αυτό είναι ένα μάθημα για το μέλλον. Να ακούμε ήδη από την πρώτη φορά ε, τις απόψεις και των δύο πλευρών. Εδώ λοιπόν δεν τίθεται το θέμα της ε, υπετιότητας, ποιος φταίει. Μας ενδιαφέρει η λύση. Και εγώ κατανοώ και την πλευρά του κράτους ε, που έκαναν τις έρευνες τους με βάση τις υποχρώσεις τους ε, και που ε, συνέκριναν ε, στοιχεία και σε άλλα αγροκτήματα όπου ίσως να μην κατέληξαν σε κάποια συγκεκριμένη άποψη. Όμως, από τον άλλο να ακούμε ότι έκανε λάθος ένα εργαστήριο, ότι εξαφανίστηκε ένα δείγμα και να λένε Λυπά, λυπούμαστε, συγγνώμη. Αυτό καταλαβαίνετε ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη μας. Μετά έρχεται και μια κρατική υπηρεσία και λέει λυπούμε θα κάναμε λάθος. Αν όμως το κάνει το λάθος αυτό ένας πολίτης απλός καταλαβαίνετε ότι θα υποστεί πολύ σοβαρές κυρώσεις. Από το πρίσμα λοιπόν του αναφέροντος αν δούμε το τι έγινε σε αυτή την μονάδα είναι λογικό να θεωρήσει ο αναφέρον ότι αυτά τα οποία υπέστη έχουν άμεση σχέση με τις εκπομπές από το εργοστάσιο. Ανεξάρτητα με το αν μπορούσε να το αποδείξει όχι. Πάντως ο ίδιο είχε υποχρέωση να προχωρήσει την όλη υπόθεση και να πάρει μια ε, καλή απάντηση. Δύσκολο μοιάζει αυτό. Προφανώ ε, ενδιαφέρεται και για αποζημίωση αν αποδειχθεί αυτό το οποίο ισχυρίζεται. Κατόπιν τούτου λόγω όλων αυτών συμφωνώ με τους ε, προραλήσαντες συναδέλφους ότι το θέμα το δει το κοινό ερευνητικό συμβούλιο και να καταθέσει μία πρόταση. Το βάρος της ε, απόδειξης δεν πρέπει να είναι στην πλευρά του αναφέροντος. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει κάποιο λόγο να ισχυρίζεται αυτά που ισχυρίζεται και πρέπει να αποζημιωθεί και ηθικά και οικονομικά είτε από το κράτος, είτε από την Επιτροπή, είτε από κάποιους θεσμούς. Αλλά αν μπείτε στη δική του τη θέση, η κτηνοτροφία κάτω από αυτές τις συνθήκες να υπάρχει ένα εργοστάσιο κοντά στο αγρόκτημα, κλείνει το εργοστάσιο, βελτιώνει την κατάσταση των ζώων, ε, λογικό δεν είναι να συμπεράνει αυτά που συνεπέρανε και νομίζω ότι ως προς αυτό θα πρέπει να δείξουμε κάποια κατανόηση. Κύριε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή για μένα ήταν προφανές από την αρχή της υποθέσεως που πάνε 10 χρόνια περίπου που εμπλέκομαι σε αυτήν και για να εξηγήσω στην Επιτροπή Αναφορών. Το αγρόκτημά μου είναι κοντά στον Ταν και εγώ από την αρχή δεν είχα καμία αμφιβολία από τα όσα έβλεπα να γίνονται στο αγρόκτημα, δηλαδή οι έρευνες που έγιναν από το Υπουργείο και από την EPA, ότι ο στόχος ήταν λάθος της έρευνας αυτής. Κατά τη δική μου γνώμη από την αρχή, αυτοί προσπάθησαν να βγάλουν τον Νταν Brennan κακό αγρότη. Εξέτασαν τα πάντα στο αγρόκτημα, προσπαθώντας να βρουν κάποιο πρόβλημα, είτε του Νταν, είτε των ζώων, είτε του του τρόπου που διαχειριζόταν το αγρόκτημά του. Ως κτηματίας, ως αγρότης, με κάποια φήμη, εγώ θεωρώ ότι ο Νταν Μπρέναν είναι εξαιρετικός αγρότης και μπορώ να φέρω και όλους τους γειτονές του εδώ, όλοι θα πούν το ίδιο ακριβώς πράγμα και δεν πρόκειται να τον προδώσουμε. Νομίζω ότι ο στόχος των διαφόρων ερευνών που έγιναν από την ε, πλευρά του κράτους είχαν στόχο να προκαλέσουν σύγχυση στα πράγματα. Επίτηδες αγνόησαν ορισμένα από τα δεδομένα τα οποία ήταν αυταπόδεικτα. Τα υψηλά επίπεδα των διαφόρων βαριών μετάλλων που βρέθηκαν στην ε, φάρμα αγνοήθηκαν ξανά και ξανά. Ένας μάλιστα από το Υπουργείο είχε πει προηγουμένως ότι μειώθηκε η παραγωγή από το 1999 του, του εργοστασίου δηλαδή και, και έληξε το 2008. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Σχετικά δηλαδή με, την μεγάλη, με τον οικοδομικό οργασμό στην Ιρλανδία. Φαντάζεστε ότι μέσα σε εκείνο το οικοδομικό οργασμό η δραστηριότητα του εργοστασίου μειωνόταν από το 99 με το 2008. Όχι δούλευαν 24 ώρες το 24 ώρες σε ορισμένες περιόδους, σε ορισμένα ε, ε, τμήματα εκείνης της περίοδου. Ναι, μειώθηκε το 2007 και μετά η δραστηριότητα του εργοστασίου ε, παραγωγής πλήνθων και το 2007 όταν άρχισε η κρίση και όταν πια εντάθηκε το 2008 σταμάτησε. Είπα και πριν ότι είδαμε τώρα δύο γερανούς γιατί ξαναρχίζει τώρα η δραστηριότητα ε, στην, ε, στο Δουβλίνο καθώς έβγαμε για το αεροδρόμιο. Υπήρχαν όμως εκατοντάδες από το, 2000, από το 1999 μέχρι το 2007. Εκεί η παραγωγή του εργοστασίου αυτού δεν είχε μειωθεί από το 1999 μέχρι το 2008. Και τα προβλήματα αυξήθηκαν ταυτόχρονα την ίδια περίοδο. Είναι εκπληκτικό να πάει να δει κανεί τώρα στο αγρόκτημα του Ντάν πόσο έχουν βελτιωθεί τα ζώα, πόσο έχουν βελτιωθεί η παραγωγή γάλακτος και δεν αδικό τον Ντάν που δεν επέτρεψε στο Υπουργείο να έλθει ξανά να ζυγίσει τα ζώα γιατί έχει εξοδεύσει περιουσίες τα τελευταία δέκα χρόνια από τις ιστορίες αυτές που επέβαλε το Υπουργείο. Επίσης για να κάνει κάθε τι που μπορούσε, δηλαδή να λαμβάνει δείγματα αίματος από τα ζώα κάθε δύο εβδομάδες, να αλλάζει τη διατροφή. Είχε δίκιο που τους ε, απελαόρευσε την είσοδο τα τελευταία δύο χρόνια. Εγώ είδα τα ζώα του πολλές φορές τα τελευταία δέκα χρόνια. Ήταν προφανές ότι κάτι τα πειράζει και τώρα αυτό έχει σταματήσει. Ακόμα και τα δέντρα του αγροκτήματος. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικό εμπειρογνώμονας για τα δέντρα για να βλέπει το 2003 και 2004 ότι κάτι τα ενοχλούσε τα ζώα. Πάτε σήμερα στο αγρόκτημά του τα δέντρα είναι υγιή, διότι το εργοστάσιο έχει κλείσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ακούοντας αυτά που είπαν ορισμένοι από αυτούς που παρενέβησαν σήμερα, είπαν ότι δεν υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις, ενώ υπήρχαν ενδείξεις μειωμένη απόδοση, μειωμένη ανάπτυξη των σώμα. Είναι απίστευτα επαγγελματίε άνθρωποι να έρχονται και να λένε τέτοια πράγματα εδώ. Εγώ έχω εδώ διαθέσιμο πλήρη κατάλογο χιλιάδων ε, δειγμάτων αίματος. Όπως είπε ο διπλανό μου, ορισμένα από τα δείγματα αυτά είχαν υπερβολικά υψηλά επίπεδα πριν να μπορέσει καν να γίνει οποιαδήποτε μόλυνση των δειγμάτων αίματος στο εργαστήριο. Και όπως είπε η κυρία ο κύριος Ευρωβουλευτής μάλλον από εγκεκριμένο εργαστήριο. Επίσης είναι δυνατόν χάθηκαν λέει δείγματα αίματος. Χάθηκαν, απολέστηκαν. Αν εγώ ως αγρότης ή ο Νταν Μπρέναν ως αγρότης κάναμε τέτοια λάθη στην καθημερινή μας διαχείριση του αγροκτήματος για οτιδήποτε υποτίθεται είμαστε υπόλογοι θα τρώγαμε πρόστιμα γερά για την πολλαπλή συμμόρφωση. Πού λοιπόν είναι το στοιχείο της δικαιοσύνης εδώ για τον μεμονωμένο αγρότη όπως την Τάν Μπρένεν. Το μόνο που θέλει είναι να προχωρήσει να αναπτύξει το αγροκτημά του, η καθημερινή του δουλειά. Και αυτά τα πράγματα του έχουν κοστίσει, να μην πω όχι μόνο χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες λιρών τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν γνωρίζω τι εννοείται με την Joint Research Committee, την μεικτή Επιτροπή Έρευνας. Γνωρίζω για την ομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά ένα πράγμα στο οποίο νομίζω πρέπει να επιμείνουμε είναι ότι ο Νταν και οι επαγγελματίε που τον βοηθούν να συμμετάσχουν στις εργασίες οποιοδήποτε σώματος ή οργάνου εγκύψει στο θέμα. Και νομίζω ότι πρέπει πράγμα το θέμα να περάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο, διότι μέχρι τώρα δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος. Νομίζω ότι η έκθεση που έχει συνταχθεί και η οποία αγνοεί επίτηδες πολλά γεγονότα θα πρέπει να αποσυρθεί. διότι πρόκειται για προσβολή προς το πρόσωπο του Νταν Μπρέναν και την οικογένειά του. Πώς είναι δυνατόν επαγγελματίες να αγνοούν γεγονότα επειδή τους βολεύει. Ο κύριος Σκρίδη διέκοψε τον εμπειρογνώμονα της Κομισιόν όταν μιλούσε για τα δεδομένα του 2006. Είχε ωστόσο δεδομένα μέχρι και το 2008 και 2009 και φαίνεται ότι και η Κομισιόν αγνοεί τα δεδομένα αυτά. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μιράντα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Είναι ένα παράδειγμα. Εγώ έχουμε από μια ε, χώρα που παράγει γαλλό, όπως και η Ιρλανδία, και πολλές φορές ε, οι διοικήσεις δεν δίνουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όταν ε, θέλουμε τελικά να θέσουμε τον ανίσχυρο απέναντι στον ισχυρό. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν σε αυτή την αναφορά πάρα πολλά στοιχεία για να αντιστηρίξουμε την αναφορά. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει διαφάνεια. Ε, δεν ε, λαμβάνονται υπόψη κάποια στοιχεία. Υπάρχουν ε, σφάλματα. Βλέπουμε ότι δεν γίνεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, αλλά από μεροληπτούντες εμπειρογνώμονες η έρευνα και αυτό που είπαν πολλοί βουλευτέ είναι εύστοχο. Και βέβαια πρέπει να λέω πόσο και τον ανθρώπινο παράγοντα. Έξι χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα για, ένα γεωργικό, για μια γεωργική εκμετάλλευση είναι πολλά χρόνια για την υγεία και του ανθρώπου και των ζώων, ιδίω όταν εδώ ο αναφέρον ε, μας φέρνει και τα στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία της απάντηση 26 Οκτωβρίου λέει ότι διαπιστώνει παραλήψεις ε, σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις. Αλλά αυτό το επιχείρημα δεν είναι αρκετό κατά την άποψή μας. Πρέπει να εμβαθύνει. Επίσης, ε, θεωρούμε ότι οι οδηγίες όταν εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη, πρέπει να γίνονται ε, να εφαρμόζονται με αυστηρό τρόπο. Και αυτό δεν έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση. Ένα άλλο επιχείρημα, το οποίο χρησιμοποίησαν εκπρόσωποι της Ιρλανδικής κυβέρνησης, είναι η αναφορά ε, στην έλλειψη ε, μετάλλων ε, από τη διατροφή και μιλά για κάποιες ε, φυσιολογικές νόσους. Τι θα πει φυσιολογική νόσος. Ποιος μπορεί να το καθορίσει καλύτερα από τον κτηνοτρόφο που ζει κάθε μέρα και βλέπει τα ζώα του και τα ταΐζει και ξέρει και πώς είναι και τι ε, τρώνε. Αυτό μου φαίνεται μεροληπτικό. Δεν επιδεικνύεται απαραίτητη αμεροληψία και αντικειμενικότητα, γι' αυτό στηρίζουμε την αναφορά αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μιράντα. δώσω τώρα στο το λόγο στην κυρία Βέρτμαν. Θα ήθελα λοιπόν ευθύ εξ αρχή ε, να σα πω το εξή. Κοίταξτε, εγώ έρχομαι από την Αυστρία. Είναι ορεινή η χώρα και εμεί έχουμε ορεινή γεωργία. Και σήμερα το γεγονός ότι πρέπει να συζητάμε για βαρέα μέταλλα και τα συναφή, αυτό και μόνο είναι φοβερό. Κοιτάξτε, εγώ ήμουνα περίπου 6-7 ετών ε, και από τότε, από τη δεκαετία του 70, είναι γνωστή οι γνωστέ επιπτώσει των βαρέων μετάλλων στην υγεία των ανθρώπων. Δεν χρειάζεται καν να διστάσω. Στηρίζω ανεπιφύλακτα τον αναφέροντα. Πιστεύω ανεπιφύλακτα ότι ε, πρέπει να μας κατατεθεί μια πραγματικά διαφανής και ανεξάρτητη έρευνα. Είναι σοκαριστικό το γεγονός το να μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο σήμερα στην Ευρώπη. Αδιανόητο. Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η κατάσταση. Προφανώς και ο αναφέρον θα πρέπει να αποζημιωθεί να του επιστραφούν οι δαπάνες του. Ασχολείται με τη Γεωργία. Εγώ δεν έχω άμεση σχέση και γνώση της Γεωργίας, αλλά πιστεύω αυτά που λένε οι υπόλοιποι. Είναι ένας καλός Γεωργός. Αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ασχολείται και αγωνιά για τα ζώα του. Όλοι μας έχουμε οικογένειες. Εμείς ε, γνωρίζουμε τα μέλη της οικογένειάς μας. Εκείνος γνωρίζει τα ζώα του, είναι η οικογένειά του. Εκείνος ξέρει κατά πόσον τα ζώα του ασθενούν ή όχι. Το να συζητάμε κάτι τέτοιο, σας παρακαλώ αγαπητή Επιτροπή, ε, σας παρακαλώ να οργανώσετε μία ανεξάρτητη έρευνα. Είναι ε, προφανές ότι πρέπει να συζητήσουμε την ε, αποζημίωση των δαπανών και επίσης το όλο θέμα να παραμείνει ανοιχτό μέχρι να διευκρινιστεί το όλο θέμα σε όλες του τις λεπτομέρειες έτσι ώστε να μην μπορεί να κάνει κανείς από εμά οποιαδήποτε περαιτέρω παρατήρηση. Πρόεδρος. Πανέρχομαι στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Άντρου και του δίνω το λόγο. Um, Για να δώσω μια απάντηση Θα... Για να δώσω μια απάντηση, ε, είμαι λίγο σε δύσκολη θέση σε σχέση με το τι μπορώ να εγγυηθώ ή να μην εγγυηθώ αυτή τη στιγμή από την Κομισιόν. Δηλαδή, αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι θα κάνουμε τις έρευνές μας, αλλά δεν μπορώ να δεσμευτώ ως προς το ότι ε, ποια υπηρεσία θα επιθεωρήσει, η Κομισιόν τι θα επιθεωρήσει κτλ. Από την ε, πλευρά και των αναφερόντων ε, και των συναδέλφων, μάλλον και των βουλευτών, βλέπω ότι υπάρχει επιθυμία να συνεχιστεί η έρευνα. Ιδίω ό,τι αφορά τα επίπεδα καδμίου ε, στα ζώα. Αυτό συνήγαγα, όχι συγκεκριμένα για το εργοστάσιο ε, κατασκευής πλήνθων. Θα δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ε, τώρα δεν ξέρω τι μπορώ εγώ να δώσω ως ε, εγγύηση και ως δέσμευση. Δεν μπορώ, δεν έχω εντολή για να δέσουμε αυτό περισσότερο αναφέρονται σε εφόσον το επιθυμούν έχουν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να εστιάσουμε για μια ακόμη φορά σε αυτά που έγιναν. Να μην ε, ξεχνάμε και τα ζώα. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ζώων υπέφεραν. Και η όλη εστίαση της έρευνας ε, των αρχών ήταν να αποδείξουν ότι δεν προκάλεσε αυτό το φαινόμενο το εργοστάσιο κατασκευής πλήνθων. Ήρθαν όμως μέλη της Επιτροπής και ήταν με τα μάτια τους και το περιβάλλον και τα ζώα που υπέφεραν. Και θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι συστάσεις στο τέλος όλων αυτών των εκθέσεων των αρχών ουσιαστικά τι λένε, δεν έφταιγε το εργοστάσιο, άρα χαίρεται. Μα αυτά τα ζώα τελικά αφέθηκαν στη μοίρα τους να υποφέρουν. Όταν έφυγαν όλοι αυτοί οι πυρογνώμονες, συνέχισε να υποφέρει ε, το ζωικό κεφάλαιο. Ευτυχώ έκλεισε το εργοστάσιο και δόξα το Θεώ βελτιώθηκε η κατάσταση και βελτιώθηκε σημαντικά στο αγρόκτημα. Όμω, ήταν εξαιρετικό γεγονό Δεν υπάρχει μικρόφωνο. Πρέπει να πιέσω το κουμπί. Λυπούμε για το πρόβλημα με το μικρόφωνο. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ, αλλά θέλω να ολοκληρώσω το εξή. Εάν γίνει ανεξάρτητη έρευνα, επιστημονική έρευνα, σας παρακαλώ, όλες τις πληροφορίες να τις διαθέσετε σε αυτό το φορέα. Γιατί υπάρχουν τεράστιες, τεράστιοι όγκοι πληροφοριών που παραγνωρίστηκαν και έμειναν εκτός αυτών των ερευνών. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά τα στοιχεία τους και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, εμείς τους στείλαμε τους ε, φακέλους... Ε, σχετικά με τις εκπομπές από το εργοστάσιο κατασκευής ε, Πλίντον που έκλεισε το Δεκέμβρη του 2008 και η... Α, έκλεισε μικρόφωνο. Συγγνώμη. 2007, τον Το Νοέμβριο του 2007 αλλά και αργότερα και το 2008 τους ε, δώσαμε στοιχεία όπου υπάρχει παραβίαση των κανονισμών για εκπομπές ε, που περιέχουν φθοριού χάλατα. Και η νέα νομοθεσία άρχισε να ισχύει το 2007. Εμείς δείξαμε παραβιάσεις και το 7 και το 8. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τοποθετήθηκε σε αυτές τις πολλαπλές παραβιάσεις. Ε, μιλάμε για περίπου 370 ε, παραβάσεις ε, των εκπομπών με φθοριούχο άλλας. Εγώ τις πήγα προσωπικά, ο ίδιος πήγα τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή και εδώ κάτι τρέχει, κάτι σημαίνει που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Θέλει κάποιος άλλος αναφέρον το λόγο. Δεν το νομίζω. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Μακαντρού να απαντήσει σε αυτό που μόλις, μόλις τώρα αναφέρθηκε. Δηλαδή, 370 ε, παραβάσεις, ε, δηλαδή αυτό προσπαθεί κάποιος να μας πείσει ότι δεν έχει σημασία, ότι δεν παίζει ρόλο. Κοιτάξτε, ε, Θέλω να ακούσω την άποψη του κυρίου Μπράνναν το αναφέροντος, όσον αφορά το θέμα της ε, σύγκρουσης ε, ανάμεσα στους ε, εμπειρογνώμονες. Αυτό πρέπει να εξεταστεί σε άλλο επίπεδο. Και καταλαβαίνω ότι έχουν τεθεί πολύ σοβαρά θέματα, αλλά θέλω να ρωτήσω τον αναφέροντα κατά πόσον συμφωνεί με αυτό που προτείνουμε, δηλαδή να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, να την παραπέμψουμε στο πλέον κατάλληλο επιστημονικό φορέα, γιατί νομίζω ότι το χρωστάμε στον κύριο Μπράνα να προχωρήσουμε, να μην ε, παραμείνουμε στάσιμοι σε αυτό το θέμα. Μετά από αυτή τη συζήτηση, θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Προτείνω να εξετάσουμε αναλυτικά όλα τα έγγραφα, τα οποία θέτουν υπόψη μας και οι δύο πλευρές, και μετά την ανάλυση των διαφόρων εκθέσεων, οι συντονιστές της Επιτροπής Αναφορών πιστεύω ότι θα είναι σε θέση να λάβουν την καλύτερη δυνατή απόφαση. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει ανεξάρτητα και αμερόληπτα, δηλαδή μέσω του κοινού Συμβουλίου Ερευνών, ε, την όλη υπόθεση. Και περνάμε στο σημείο 16 της μερίσιας διάταξης έξι αναφορές ε, οι οποίες αφορούν ε, την προστασία των αποδημητικών πτηνών στην Ιταλία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία και στην Ιρλανδία. 798 του 2004, 334 του 2005, 886 του 2005, 530 του 2006, 1091 του 2007, και 1374 του 2010. Ο αναφέρον είναι παρόν. Jean-Claude Domo λέγεται και εκπροσωπεί τη Βελγική Βασιλική Εταιρεία την Προστασία των Πτηνών. Κυρία Πρόεδρε, το 2005 195.000 υπογραφές ε, συνέλεξε η αναφορά μας, πολλές και από τη Μάλτα. Και στόχος μας είναι να εφαρμοστεί νομοθεσία από τη Μάλτα. Το 2005 και μετά δεν άλλαξε τίποτα. Μιλούσαμε για μια μεταβατική περίοδο που χορηγήθηκε στη Μάλτα για να προσαρμοστεί στην νομοθεσία αυτή. για το 2008, έχουμε φτάσει το 2012, η πρώτη ετήσια έκθεση το 2005 σε ό,τι αφορά ε, την υλοποίηση των δεσμεύσεων της μεταβατικής περίοδου, όπου να είναι θα ολοκληρωθεί, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει τίποτα προς το παρόν. Άρα, ποιο κοροϊδεύει ποιον. Η Μάλτα τελικά φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση να πάψει ε, η θανάτωση των αποδημητικών πτηνών, καθυστερεί με τις προθεσμίες, κερδίζει χρόνο ώστε να ικανοποιεί ε, τους κυνηγού. Και δεν εξοντώνει μόνο ε, η θαγενή πτηνά, αλλά και πολλά αποδημητικά πτηνά που είναι κληρονομιά ολόκληρης της Ευρώπης και με ποιο δικαίωμα μπορεί μια χώρα να καταπατά τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να καταστρέφει το κοινό αυτό αγαθό, να καταστρέφει σημαντικά στοιχεία της βιοπικιλότητας της Ευρώπης. Η Βελγική Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πάρα πολύ αποφασιστική απέναντι στη Μάλτα, ώστε τελικά η Μάλτα να σεβαστεί τι υποχρεώσει και τι δεσμεύσει τη. Να σεβαστεί τα πτηνά, να σεβαστεί το περιβάλλον μα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Πέτερ Κόλλο από την Επιτροπή. Thank Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ε, αυτό το θέμα νομίζουμε ότι ε, ρυθμίζεται μέσα στο πλαίσιο ε, που έχει καθορίσει η Μάλτα και το να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα εντάσσεται μέσα στις ε, γενικότερες ε, αναφορές που εξετάζουμε. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι εδώ πρέπει να συμμορφωθούμε με την απόφαση του δικαστηρίου του 2009 που καταδίκασε την Μάλτα ε, για την πρακτική που ακολούθησε από το 4 μέχρι το 2007. Και όσον αφορά το να ανοίξει και εκ νέου η εποχή αυτή του κυνηγιού, θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή έχει ενημερωθεί ότι οι αρχές της Μάλτας θα ακολουθήσουν τους ε, κανόνες αυτά που προβλέπονται στην νομοθεσία πλαίσιο. Επίσης είναι δυνατόν ε, εφέτος ε, να παρακολουθούν οι αρχές την περίοδο του κυνηγιού Αναφέρομαι κυρίως στο έναν επιστημονικό φορέα τη Θα ήθελα επίση να σα υπενθυμίσω ότι η απόφαση του δικαστηρίου του 2009 αφήνει ανοιχτή, ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι υπάρχει μια σύντομη περίοδο κυνηγιού στην Μάλτα υπό την προπόθεση βέβαια ότι καλύπτονται όλε οι προποθέσει τη ε, οδηγία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για τη Μάλτα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι πέρυσι η Μάλτα προσπάθησε να εφαρμόσει την οδηγία αλλά υπάρχει και περαιτέρω περιθώριο. Επίσης, ε, θέλουμε η Μάλτα να συνεχίσει τις ε, προσπάθειές της, ε, έτσι ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται να ληφθούν με αξιοπιστία. Όσον αφορά τώρα την παγίδευση των τεινών στη Μάλτα, θέλω να σας πω ότι πέρυσι αποφασίσαμε να παραπέμψουμε την Μάλτα σε διαδικασία επιπαραλήψη η Μάλτα από το 2004 είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ε, τηρεί τις ε, προδιαγραφές και την οδηγία για το κυνήγι των πτηνών. Η ε, Μάλτα βέβαια τώρα πλέον επιτρέπει, η πέρυσι επέτρεψε μόνο ένα είδος να είναι αντικείμενο κυνηγιού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε το Φεβρουάριο αυτού του έτους να συνεχίσει αυτή τη διαδικασία επιπαραλήψη με βάση το σχετικό άρθρο της ε, Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να επενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς ε, της διαδικασίας που ακολουθούνται στη Μάλτα ε, και για να διαπιστωθεί κατά πόσον η Μάλτα τηρεί τις προδιαγραφές που αναφέρονται για το κυνήγι στη χώρα σας ευχαριστώ. Παρεμβάσεις. Η ομάδα μας, κυρία Πρόεδρε, επιθυμεί η αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή. Βεβαίω, η παραπομπή στην ε, προσφυγή της Επιτροπής δείχνει ότι ο φάκελος δεν έχει κλείσει. Επανέρχομαι στην εφαρμογή της οδηγίας για τη βιοπικιλότητα. Οι χώρες μέλη νομίζω δεν δείχνουν επαρκές ενδιαφέρον. Τα παίρνουν τα πράγματα αυτά πολύ ελαφρά και αυτό είναι προφανές στην περίπτωση της Μάλτας. Το κυνήγι συνεχίζεται, χιλιάδες πτηνά θανατώνονται, θέλουμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρε, αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, τότε θεωρώ ότι η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και να, την, να παρακολουθούμε τη συνέχεια. Το 17 τώρα, η αναφορά 1518 του 2008, 997 του 2007 και 1503-07. Πρόκειται και οι τρεις έχουν αντικείμενο την προστασία των πουλιών στην Βουλγαρία. Είναι παρούσα η κυρία Ειρήνα Ματέβα, εξ ονόματος της Βουλγαρικής Εταιρείας για την Προστασία των Πουλιών. Έχετε το λόγο. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με προσκαλείτε τώρα για δεύτερη φορά ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών. Θα μιλήσω με λίγα λόγια για την ε, αναφορά 1518 του 2008 και την 997 του 2007 και θα ήθελα να σας πω καλά νέα για τις δύο αυτές αναφορές. Θα ήθελα, όπως ε, είπα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ, διότι η κατάσταση, η κατάσταση σχετικά, ε, η κατάσταση στην οποία αναφέρονται οι δύο αυτές αναφορές δεν βελτιώνεται. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις χειροτερεύει. Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό τόπων Natura 2000 για τα πουλιά, θα ήθελα να πω ότι εξακολουθούμε να μην έχουμε εγκεκριμένες ε, περιοχές ειδικής προστασίας. Οι περισσότερες από αυτές είναι στις ακτές της ε, Μαύρης Θάλασσας και τις θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ήδη οριστήσεις περιοχές. Στην πραγματικότητα όμως σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία δεν είναι. Εκτός από αυτό έχουμε ε, περιοχές ειδικής προστασίας που ακόμα δεν έχουν οριστεί για λόγους οικονομικούς και μία από τις περιοχές αυτές είναι η Ρίλα, σημαντική περιοχή στο, στη νότιο-δυτική Βουλγαρία και αυτό διότι εκεί ε, είναι πολλά έργα χιονοδρομικών κέντρων και το άλλο είναι στην Καλιάκρα όπου εκεί δημιουργείται αιωλικό πάρκο θα σας πω σε λίγο. Παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλουμε και εμείς αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δύο περιοχές αυτές δεν υπάρχει σχεδόν καμία ελπίδα να οριστούν ως περιοχές Natura 2000 εάν δεν αναλυφθεί δράση. Και σχετικά με την περιοχή δικής προστασίας Καλλιάκρα και την 1518 το αιωλικό πάρκο που κατασκευάζεται στην Ντόμπρουτζη έχει όλο και περισσότερες επιπτώσεις και μέχρι τώρα έχουμε 3.928 ανεμογεννήτριες που έχει εγκριθεί η εγκατάστασή τους και προχωρεί πολύ γρήγορα το αιωλικό αυτό πάρκο και μάλιστα τους τελευταίους μήνες η έγκριση εγκατάστασης νέων αιωλικών πάρκων επιταχύνεται διαρκώς. Από όλη αυτή την ταχύτατη εξέλιξη σε μικρά μέρη της Βουλγαρίας στην περιοχή της Ντόμπρουτζε αυτά πλήττουν τα αποδημητικά είδη πουλιών, ένα είδος χήνας, δηλαδή που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει, είναι απειλούμενο είδος παγκοσμίω και που αυτά κινδυνεύει να χαθεί όλος ο πληθυσμός των πουλιών αυτών στην περιοχή του Ντόμπρουτζε. Και λόγω της λειτουργίας των αιωλικών πάρκων στην Καλλιάκρα διαπιστώνουμε ήδη τη ζημιά που έχει υποστεί το είδος διότι χάνεται ο βιότοπος όπου ε, κινούνται και ψάχνουν τροφή. Οι χήνες αυτές δεν, δεν έρχονται πλέον στους βιοτόπους αυτούς και χάνονται οι βιότοποι αυτή της Καλιάκρα. Εκτός από αυτό, μόλις πριν από ένα μήνα διαπιστώσαμε ότι το αιωλικό πάρκο της Καλιάκρα που το θεώρησε η βουλγαρική κυβέρνηση ως μεγάλη επιτυχία ότι δεν θα κατασκευαστεί καθόλου. Επιστώσαμε λοιπόν ότι έχει αρχίσει η κατασκευή αυτού του ολικού πάρκου και τελικώ αυτό θα γίνει, θα υλοποιηθεί στην περιοχή αυτή. Και τώρα εκτός από αυτό η ανάπτυξη των αιωλικών πάρκων στην περιοχή αυτή αρχίζει και απειλεί και άλλες περιοχές πολύ σημαντικές για σημαντικές για την Χίνα διότι μεγάλα αιωλικά πάρκα εγκρίθηκαν και μάλιστα χρησιμοποιούν προκαταρκτικές άδειες για να αποφύγουν τη διαδικασία του υπερτέρου δημοσίου συμφέροντος. Έτσι λοιπόν, απαιτείται άμεση αντίδραση. Αντίδραση που να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη, αλλιώς θα χαθούν αυτοί οι βιότοποι για πάντα. Ζητούμε να οριστούν οι περιοχές Ρίλα και Καλλιάκρα ως περιοχές Natura 2000 το δυνατόν συντομότερο και οι διαδικασίες αυτές να λάβουν προτεραιότητα και να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την κατεύθυνση της αιτιολογημένης γνώμης για παραβίαση από πλευρά της βουλγαρικής κυβέρνησης και η δική σας Επιτροπή Αναφορών να ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει πίεση με τη σειρά της στη βουλγαρική κυβέρνηση να σεβαστεί τις διατάξεις της οδηγίας για την προστασία των πουλιών. εκπρόσωπος Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προβλήματα με τον ορισμό των ε, τόπων Natura 2000 στην ε, Βουλγαρία και θέλω να ευχαριστήσω ε, τους αναφέροντες για τις πληροφορίες που μας έδωσαν, καθώς και τους βουλευτές, τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών που εκ των προτέρων δραστηριοποιήθηκαν και έκαναν ε, και το 2010 τον Ιούνιο τη διερευνητική αυτή επίσκεψη στη Βουλγαρία. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν τεθεί, θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διάλογο με διαφόρους πολίτες, με κυβερνικές οργανώσεις και λαμβάνουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα θέματα. Επίση, έχουμε διάλογο και με τις εθνικέ αρχές και συνεχώς ζητούμε πληροφορίες από αυτές για τον ορισμό των ε, ειδικών ζωνών προστασία, ε, καθώς ε, και στοιχεία για τις άδειες δόμησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα τα οποία προβλέπονται και από τις συνθήκε της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την αποτελεσματική προστασία των ειδικών ζώνων προστασίας και τον ε, ορισμό τους βάσει τη νομοθεσία ό,τι αφορά τον ορισμό των ειδικών ζώνων προστασία. Θα ήθελα επίση να σα αναφέρω ότι λόγω αυτού του διαλόγου και της, ε, των διαδικασιών επιπαραβάσεις που έχουν κινηθεί, έχουμε επιτύχει διάφορα πράγματα, τα οποία θα ήθελα να σας αναφέρω. Το Μάιο του 2011, οι Εθνικές Αρχές έλαβαν απόφαση για επέκταση του δικτύου ζωνών ειδικής προστασίας στη Βουλγαρία. Πάνω από 244.000 εκτάρια καλύπτει αυτή η ζώνη στη Βουλγαρία. Και η διαδικασία κινείται με καλούς ρυθμούς για τη Δυτική Ροδόπη και για μια περιοχή στα Πυρηναία. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τι ε, ζώνε Προστασίας προστασία, υπάρχουν κάποια άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε στι αρχέ Μαΐου με τις ε, βουλγαρικές αρχές. τι βουλγαρικέ αρχέ. Ό,τι αφορά την Καλλιάκρα, θα θέλαμε να ενημερώσουμε την αναφέρουσα αλλά και την Επιτροπή Αναφορών ότι υπήρξε μια έγγραφη προεδοποίηση, μια επιστολή που εστάλει το Σεπτέμβριο του 2011 στις βουλγαρικές αρχές. Εκεί μιλούμε για την ανεπαρκία της όλης διαδικασίας ε, και επίσης ε, συζητούμε και αυτό το περιβαλλοντικό έργο το οποίο έθεσε και η αναφέρουσα. Οι υπηρεσίε τη Κομισιόν αξιολογούν τα πράγματα. Θέλω να, να διαβεβαιώσω και την αναφέρουσα και τα μέλη τη Επιτροπή σα ότι οι υπηρεσίε τη Κομισιόν θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση και εφόσον αυτό χρειαστεί, προβλέπουν οι συνθήκε και συγκεκριμένα το άρθρο 258, περαιτέρω ενέργειες τις οποίες και θα λάβουμε, ε, τις οποίες και θα προβούμε για να προστατεύσουμε το, τη φύση στην Βουλγαρία. Ευχαριστούμε πολύ την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος θέλει το λόγο, η κυρία Μιράντα. Νομίζω ότι αν κανείς άλλος δεν θέλει το λόγο, ε, θα ήταν σωστό να πάρω το λόγο για να στηρίξω την αναφορά. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω την αναφέρουσα για να πω ότι είναι σωστή η αναφορά, γιατί μου θυμίζει και πολύ αυτά που γίνονται στη δική μου χώρα, που δεν ορίζονται σωστά οι ζώνες της προστασίας. Οι κυβερνήσεις τελικά, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κινούνται μόνο ε, με βάση κάποιες διαδικασίες επί παραβάση και όχι από μόνες τους. Δεν αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία από μόνες τους, ενώ θα έπρεπε να έχουν επίγνωση είναι σημαντικό να έχουν αυτές τις ζώνες ειδικής προστασίας και αυτό, αυτό δικαίως, όχι μετά από μια διαδικασία ε, επί παραβάση ή επειδή θα τους επιβληθεί κάποιο πρόστιμο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι σημαντική η αναφορά αυτή η ανεπάρκεια αυτή με τους ορισμούς ε, φαίνεται ότι θα διορθωθεί τελικά από την βουλγαρική κυβέρνηση και επειδή υπάρχουν και όλες αυτές οι διαδικασίες σε παραβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με όλα αυτά τα ολικά πάρκα ε, και με όλα αυτά τα έργα που δεν ελέγχονται καθόλου αυτό που τελικά βλέπουμε είναι ότι χάνονται οι κότοποι, χάνονται οικοσυστήματα. Εμείς πιστεύουμε από τη δική μας πολιτική ομάδα ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να γίνει στο δυνατόν πιο γρήγορα η σχετική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Ε, μετά από αυτή τη συζήτηση, λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές οι αναφορές. Η Επιτροπή Αναφορών ε, θα παρακολουθεί στην υπόθεση, πάντοτε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και περνάμε στο τελευταίο σήμερα διάταξης για σήμερα, που είναι η αναφορά 1044 2011 αναφορά της Τζοάννα Σουέιμπ αφορά το εμπόριο προϊόντων φώκιας. Η αναφέρουσα είναι στην αίθουσα και θα μας κάνει μία παρουσίαση σε PowerPoint. Μινούτε. Περιμένουμε ένα-δύο λεπτά για να δούμε τις διαφάνειες. Um, ε, ευχαριστώ. Εκπροσωπώ την Humane Society International και 20.000 ε, πολίτες οι οποίοι έχουν συνυπογράψει την αναφορά από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ λοιπόν την ε, πρόεδρό σας κυρία Μπασέσκου η οποία μας επιτρέπει να προσέλθουμε εδώ ενώπιόν σας για να εξηγήσουμε την αναφορά μας για την Συμφωνία ΣΕΤΑ και την προσφυγή του Καναδά στον Οργανισμό ε, Παγκόσμιο Οργανισμό εμπορίου. Το Μάιο του 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία ε, ψήφισε υπέρ μιας απαγόρευσης του εμπορίου προϊόντων φώκιας μετά από δεκάδες ευρύτατη συζήτηση για την, το εμπόριο ε, από αυτό το σκληρό κυνήγι. Θα ήθελα να σας θυμίσω οπτικά τώρα πώς αποκτώνται αυτά τα προϊόντα φώκιας. θα χρειαστώ μια τεχνική βοήθεια. Okay. That will go. Okay. Να λοιπόν μπορείτε τώρα να δείτε αυτό το φιλμ. Να σας δείξουμε τώρα ένα σύντομο φιλμ από το κυνήγι της περσινής χρονιάς. Ο Καναδάς ισχυρίζεται ότι το κυνήγι της φώκιας γίνεται με ε, κατάλληλο, με ανθρώπινο τρόπο εντό εισαγωγικών. Εμείς μιλούμε για σφαγή. Δεν είναι μονάχα ένα παράδειγμα για το πώς οι καναδικοί κανονισμοί δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν την απάνθρωπη αυτή φύση του κυνηγιού της φώκιας, αλλά ο ίδιος ο Καναδάς δεν επιβάλλει την τήρηση των ε, κανονισμών αυτών. Είδαμε και πέρσι πάλι η ομάδα μας δηλαδή ε, έβγαλε ταινία ε, νεογνά της φώκιας τα οποία καρφώνονται ζωντανά σε γάτζους και τα τραβούν πάνω στο χιόνι και άλλες ε, ε, σκηνές όπως θνίσκοντα νεογνά φώκιας τα οποία φωνάζουν πάνω σε σωρούς πτωμάτων άλλων μικρών και φώκες τις οποίες πυροβολούν κατ' επανάληψη στα ανοιχτά νερά. Όλα αυτά είναι προκαλούν έντονα ε, αρνητικά συναισθήματα αλλά χάρη τουλάχιστον στην απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων φώκιας χιλιάδες φώκες γλίτωσαν. Πέρσι ε, φωνεύτηκαν μόνο 38.000 ε, φώκες του είδους του Harp Seal ενώ ο αριθμός είχε φτάσει 350.000 πριν από 5 χρόνια. Έχει μειωθεί λοιπόν η σφαγή αυτή ως απόρρια της απαγόρευσης ε, του εμπορίου στην ε, Ευρώπη. Το ίδιο πριν από λίγους μήνες η Ρωσία απειγόρευσε την εισαγωγή και εξαγωγή ε, προϊόντων φώκιας, δηλαδή δερμάτων γουναρικών και υπάρχουν τώρα σημαντικές εμφωλίες και μεταξύ των Καναδών εάν θα βρεθούν έμποροι να αγοράσουν τα προϊόντα αυτά αφού ήδη τα αποθέματα γουναρικών που έχουν μένουν απόλυτα. Ο Καναδάς βέβαια είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένος με την ευρωπαϊκή αυτή απαγόρευση. Μετά από πολλούς μήνες ε, που απειλούσε τελικά ζήτησε, προσέφηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και ζήτησε ένα dispute panel να ανοίξει. Εμείς οι αναφερόμενοι θεωρούμε ότι αυτή η προσφυγή ενώπιον του ΠΟΕ δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απευθείας επίθεση κατά των ηθικών αξιών των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των δημοκρατικών τους διαδικασιών. Δεν υπάρχει ουδέμια αμφιβολία βεβαίως ότι οι δικηγόροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υπερασπιστούν τον κανονισμό ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου εφόσον φτάσει εκεί. Ωστόσο εμείς ως Ευρωπαίοι πολίτες αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται ε, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την καναδική κυβέρνηση χωρί να έχει βάλει ω όρο την απόσυρση τη προσφυγή στον ΠΟΕ για να μπορέσουν να γίνουν αυτέ οι διαπραγματεύσει. Είναι απαράδεκτο να συνεχίζει τη διαπραγμάτευση αυτή τη συμφωνία, ενώ ταυτόχρονα ο Καναδά κάνει ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει το δικαίωμα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να αποφασίσει δημοκρατικά ποια προϊόντα θέλει να επιτρέψει να εισάγονται στην επικράτειά τη. Μα ικανοποιεί το γεγονό ότι ε, ψηφίστηκε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εμπορικές σχέσεις με τον Καναδά πέρσι και που θεωρεί ότι δεν πρέπει να, να γίνει η συμφωνία αυτή, αλλά το πρόβλημα της φώκιας εξακολουθεί να είναι, όπως λέμε στα αγγλικά, ο ελέφαντας μέσα στο συνέθουσα που δεν, ε, που δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς. Γι' αυτό με την αναφορά μας ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να υπεραμεινθεί της ίδιας του της νομοθεσίας και να μην υποστηρίξει την συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά, μέχρι ότου αυτό αποσύρει την προσφυγή του στον ΠΟΕ. Α μην λησμονούμε επίση ότι εδώ διακυβεύονται πολύ περισσότερα πράγματα από ότι η απλή απαγόρευση ε, κυκλοφορία ε, προϊόντων φώκια. Πρόκειται για την ίδια την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Εάν το Κοινοβούλιο δεν υπεραμεινθεί της ίδιας του τη νομοθεσία, οι απλοί πολίτες όπως εγώ, όπως και άλλοι 20.000 που έχουν υπογράψει την ε, αναφορά, θα χάσουμε κάθε εμπιστοσύνη στην πολιτική διαδικασία. Πώς εμείς ως πολίτες υποτίθεται ότι θα εμπιστευόμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν αυτό δεν στηρίξει με έντονο τρόπο την νομοθεσία την οποία έχει και αυτό ψηφίσει. Διοχητεύοντας έτσι εκατομμύρια σε μια χώρα η οποία δεν σέβεται τις ηθικές μας αξίες. Με την κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να το πράξει αυτό και εμείς ζητούμε να προχωρήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις αυτές. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Well, uh, thank you very much, Madam Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ε, και ευχαριστώ και τους ε, αναφέροντες ε, είναι αλήθεια ότι ο Καναδάς ε, ζήτησε να υπάρξει ε, μια διαδικασία διευθέτησης και διαιτησίας. Αυτό έγινε το Φεβρουάριο του 2011 και το Μάρτιο ενώσαμε τις δυνάμεις μας. Η διαδικασία στη Γενέβη είναι στη φάση που θα συσταθεί το πάνελ και το πάνελ θα εξετάσει τους ισχυρισμούς τόσο του Καναδά όσο και της Νορβηγίας. Εμείς πιστεύουμε αυτή η απαγόρευση με τους κανόνες του ΠΟΕ ε, και δεν είναι προστατευτική η οδηγία, αλλά πρέπει πραγματικά ε, να ανταποκριθεί ε, στις ανησυχίες περί των Ευρωπαίων πολιτών. Και κατόπιν τούτου δεν, είναι, δεν ασκεί διακριτική μεταχείριση η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προστατεύσει, θα υπεραμεινθεί τις θέσεις της στη Γενέβη. <clears throat> Τώρα, αυτά σε σχέση με την απαγόρευση ε, κυνηγιού της φώκιας, αυτό δεν είναι σωστό. Κάτι τέτοιο δεν θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κάθε μέλος του ΠΟΕ έχει το δικαίωμα να καταφεύγει σε διαδικασία διαιτησίας εφόσον πιστεύει ότι παραβιάζουν οι συμφωνίες του ΠΟΕ. Ο Καναδάς κατέφυγε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι απόλυτα συμβατό με την, τους νόμους του ΠΟΕ, ακόμα και αν πιστεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σέβεται τους κανόνες του ΠΟΕ. Το όλο σκεπτικό πίσω από τη διαιτησία είναι να προσφέρεται στα κράτη-μέλη ένα νομικό πλαίσιο για να επιλύονται οι διαφωνίες. Τώρα, αν ένα μέλος δεν συμφωνεί με τις συστάσεις ε, του ΠΟΕ, τότε πρέπει να επιβάλλονται ε, κυρώσεις ε, και ενδέχεται προφανώς να επιβάλλονται κυρώσεις. Τα μέλη του ΠΟΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορούν να καταφύγουν σε ένα τέτοιο μηχανισμό παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έκανε ποτέ πριν να εξαντλήσει όλες τις άλλες δυνατότητες να εξευρεθεί λύση. Το σύστημα βοήθησε ε, στο να αποφευχθούν πόλεμοι εμπορικοί, ο μηχανισμός προστατεύει τα αδύναμα μέλη από τα πιο ισχυρά. Η παρέμβαση σε αυτή τη διαδικασία ε, μπορεί να οδηγήσει τον Καναδά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό ε, θα ήταν επιζήμιο για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου υπάρχει συμφωνία και ε, ανάμεσα στον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην προκληθούν εμπόδια στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και ενδέχεται να γνωρίζετε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις διαπραγματεύσεις δεν τις συνήρτησε με το να ε, σταματήσει ο Καναδάς ε, τις ε, προκλήσεις που προβάλλει στον ΠΟΕ. Η εμπορική συμφωνία Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν εφαρμοστεί, θα συνεπάγεται σημαντικά οικονομικά ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Και επίσης θα περιλαμβάνει και κεφάλαια που θα έχουν σχέση με την αηφόρο ανάπτυξη, κάτι που μακροπρόθεσμα είναι χρήσιμο ε, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον Καναδά, κυρίως βέβαια για τον ε, Καναδά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Τέιλορ τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώ τους Πρασίνους. Είμαι μέλλον ε, της Διεθνούς Εμπορικής Επιτροπής και πραγματικά ανησυχώ ιδιαίτερα για το ότι η Κομισιόν φαίνεται ανίσχυρη να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ρητός εξέφρασε τις ανησυχίες του το Μάιο του 2009. Είχα πολλέ συνομιλίε και στο πλαίσιο της Διεθνούς Εμπορικής Επιτροπής και όχι μόνο για τις φώκες. αλλά και για πολλά άλλα είδη και για τις αμμώδεις ε, ποιήσεις και για τις άρσεις, ε, για, για τις εξαιρέσεις από τη θεώρηση κτλ. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Έχουμε αυτή την ε, ρύθμιση ΣΕΤΑ Πώς μπορεί κανείς να την υποστήριξει. Βλέπουμε επίσης ε, μια πράξη εχθροπραξίας, αν θέλετε, από τον Καναδά που χρησιμοποιεί ε, τον ΠΟΕ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι είναι αυτό ε, κρίμα και ντροπή. Πρέπει να μας δώσει μια εξήγηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να προσπαθήσει να διασκεδάσει τουλάχιστον την εντύπωση που έχουμε εμεί δημιουργήσει. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σκίνερ, λέει πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, φυσικά για πολλούς από εμάς που ασχοληθήκαμε και κατά το παρελθόν με εξοδαφικά ζητήματα και τον Καναδά και θυμάμαι πολύ καλά όταν έλαβε μια απόφαση για τον αμίαντο ο ΠΟΕ δεν φαίνεται να έχει περάσει και τόσο ε, καιρό από τότε. Ήταν το πρώτο κοινωνικό νομοθέτημα τελικά, ε, το οποίο πέρασε με έφεση στον ΠΟΕ διότι αποδείχθηκε ότι αφορά τις ζωές ε, πάρα πολλών. Αυτή η διαφορά φαίνεται να είναι μεταξύ Κομισιόν και Καναδά, αλλά τελικά πάρα πολλοί άνθρωποι θίγονται. Το θέμα της θανάτωσης, ε, της φαγής ε, των φωκιών και της χρήσης του δέρματός τους είναι ένα θέμα που φύγει και αφορά πάρα πολλούς. Και στη δική μου περιφέρεια έχω συναντηθεί με πάρα πολλούς πολίτες που πραγματικά ε, έχουν κάποιες ελπίδες σε σχέση με αυτά τα οποία ζητά η Κομισιό. Και αυτά θα γίνουν με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ε, θα κριθεί απαραίτητο. Εγώ γνωρίζω τους ε, νομικούς περισμούς των ΠΟΕ, αλλά έχουν δοκιμαστεί κατά το παρελθόν. Πρέπει να έχουμε κατά νου τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά και πρέπει να υπάρχει και κάποια ευελιξία. Να περιμένουμε βέβαια να οι συζητήσεις γιατί αλλιώς ε, θα φανούμε πάρα πολύ αδύναμοι ευθύς εξ αρχής. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχουν ικανοποιητικά επιχειρήματα ε, γιατί υπάρχουν και πολλοί άλλοι ανθρώπινοι λόγοι που μπορούν να προβληθούν. Δεν είμαι δικηγόρος, αλλά μπορώ να πω στην Επιτροπή ότι ορισμένα πράγματα γίνονται, ε, παρότι παλαιότερα μας έλεγαν ότι δεν μπορούν να γίνουν σε σχέση με τον ΠΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Η αναφερόμενη πως επιθυμεί να προσθέσει κάτι ή κάποιο από τους άλλους παρισταμένους. Δεν έχει μικρόφωνο η πρόεδρος. Μα σκουζάτε, στην κλούζια τη κουτσέιδα, θα σα πω η κλούζια Προτείνω να στείλουμε επιστολή στον ε, Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για τις εμπορικές σχέσεις για το θέμα αυτό. Ουδής άλλος επιθυμεί να λάβει το λόγο. Έχουμε εξαντλήσει επομένως τα θέματα της ημερησίας διατάξεως για σήμερα. Η κυρία Μιράντα. Με συγχωρείτε βέβαια, επιμένω κάπως. Μήπως μπορούμε να δούμε την αναφορά υπαριθμών 37. που αναμένει απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν είναι δυνατόν κυρία Πρόεδρε. Am uh, Σημειώνουμε το αίτημά σα. Η γραμματεία έχει λάβει το αίτημα να κρατήσει ανοιχτή ανοιχτές μάλλον τις αναφορές 37 και 38 όπως είπατε αν υπάρχει συνάδελφος που θέλει να ανοίξει αναφορά της λίστας Β όχι σας ευχαριστώ λοιπόν για την συμμετοχή σας η επόμενη συνεδρίασή μας θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου. Εδώ λήγουν οι εργασίες.